Okay. Χαίρετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πέρασε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ήταν υπεραρκετό. Και ξεκινούμε με μια σειρά από προτάσεις που αφορούν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις συνέπειες της ένταξης αυτής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δεν έχουμε παρόντες όλους τους εισηγητές μας και γι' αυτό το λόγο προτείνω να ξεκινήσουμε με την Επιτροπή πρώτα που μας κάνει την παρουσίαση και με την αλλαγή αυτή να αφήσουμε και ένα χρονικό περιθώριο στους εισηγητές μας ώστε να έρθουν για να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Είναι η Επιτροπή παρούσα. κύριος Ντεβινιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ξέρετε, έχουμε τέσσερις ε, συμφωνίες πέραν των ε, γενικών ε, δεσμεύσεων και των διαπραγματεύσεων στις οποίες έχει διαδραματεύσει ηγετικό ρόλο, η, διαδραματίσει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στις από 15 χρόνια. Τέσσερις συμφωνίες που καλύπτουν τέσσερις σημαντικούς για μας τομείς. που προχωρούν μέσω ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Η πρώτη αφορά τον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων και αφορά την, ε, το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. Όπως θα ξέρετε έχουμε συμφωνήσει με τους Ρώσους ότι μπορούν να διατηρήσουν το σύστημα προστασίας, όχι όμως ακριβώς προστασίας υποχρεωτικών ε, μέτρων επενδύσεων στο ιστορικό της Ρωσίας που, ήταν, ε, που είχαν κριθεί ε, ασυμβίβαστα με το TRIMS, με, το, με τη συμφωνία δηλαδή τη σχετική με τα μέτρα άμεσων επενδύσεων ενώ του 2018 που υποχρέωναν την Ρωσία να σταματήσει τις, ε, τα μέτρα που αντιβαίνουν στην ε, ελευθερία ε, μετακίνησης επιχειρήσεων και έτσι έχουμε αυτή τη συμφωνία για όγκο 900 εκατομμυρίων για τις μηχανές και 8,2 δις για τα συστατικά και τα ανταλλακτικά. Το επίπεδο των εξαγωγών λοιπόν για το 2010 παρά τα μέτρα επενδύσεων της ρωσικής ε, ε, κυβερνήσεως διατηρούνται όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος είναι η εισαγωγή μιας ποσόστοσης απαλλαγμένης από τελωνιακούς δασμούς για επίπεδα χαμηλότερα αυτών του 2010. Ποσόστοση λοιπόν αδασμολόγητου αντί για διαφορετικές, ε, διαφορετικά ποσοστά αδασμολόγητου που κειμενόταν μεταξύ του 5% και του 10%. Τώρα δεν αφορά τα, τις εξαγωγές σε είδη ξυλίας. για την ε, χαρτοβιομηχανία και για την επιπλοπία ε, συγκεκριμένα με τη δυνατότητα για εξαγωγή με χαμηλότερους δασμούς, 13 και 15% αντίστοιχα για τα δύο είδη ξυλίας, αντί για το, 25% που επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ρωσική Κυβέρνηση Σιλίβδιν. Ένα σύστημα μάλιστα με μια επιτροπή, τη λεγόμενη επιτροπή ξύλου, ξυλίας, που θα διαχειρίζεται τα θέματα αυτά και προσδιορισμό για ...30% για τις νέες αγόμενες επιχειρήσεις, νέες αγόμενες στο σύστημα. Έχουμε επίσης ένα μακροσκελή κατάλογο πρώτων υλών στις ε, δεσμεύσεις γενικά της Ρωσικής ε, Ομοσπονδίας Ενόμψη της Προσχώρησης, το ΟΜΠΕ, και έχουμε πει ότι αν θέλει η Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει για τις ε, πρώτες αυτές την τον εξαγωγικό δασμό, μπορεί με δύο μήνες περιθώριο προαγγελία, προαναγγελία να το πράξει. τελευταία συμφωνία αφορά τις υπηρεσίες. Και εδώ εξασφαλίσαμε ότι διμερεί συμφέροντα ε, που προκύπτουν από τις σχέσεις μας, από τις συμφωνίες μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία διαφυλάσσονται στον τομέα των θαλασσιών μεταφορών αφενός με ειδική μεταχείριση για τις ε, ναυτιλιακές εταιρείε και για την απασχόληση προσωπικού όπως συμφωνήσαμε την δυνατότητα για μετακίνηση προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών. Δυνάμει της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε στους εισηγητές. Όπως σας είπα υπάρχουν τρεις εισηγητές για τα τέσσερα αρχαία. Παύλ Ζαλεύσκη είναι εισηγητή ε, τη Συμφωνία ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία σχετικά με το εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. Ένα από τα τέσσερα αρχεία τα οποία μα παρουσίασε η Κομισιόν. Παύλ Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό που διαπραγματευτήκαμε επιτέλους αυτή τη συμφωνία, την πρόσβαση της Ρωσίας στον ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, ε, συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται το εμπόριο γενικότερα στον κόσμο αλλά και για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας δημιουργεί ένα μηχανισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση των εξαγωγών ε, ε, μερών μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου η Ρωσία κατάφερε η Ρωσία να διαφυλάξει το πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα των αυτοκινήτων ε, στην παραγωγή εξαρτημάτων και μερών μηχανοκινητών οχημάτων είναι όλο και πιο αυστηρές ε, οι συνθήκες πόλης αυτοκινητών στην ρωσική αγορά. Αυτά τα μέτρα, ωστόσο, ε, δεν είναι σύμβατα. Είναι μέτρα επενδυτικά που δεν είναι σύμβατα με τον ΠΟΕ. Θα συνεχίσουν ωστόσο έως το 2011. Έτσι λοιπόν ο λανθάνων φόβος είναι ότι οι πολιτικές συνέπειες ε, ε, αυτής της προσπάθειας προοδευτικής απελευθέρωσης ε, του τομέα των αυτοκινήτων στην Ρωσία θα αντισταθμιστεί από τις συνέπειες αυτού του TRIPS. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό διασφάλισης της κατάστασης των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολύ σημαντικό Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, ειδικότερα όταν μελετάμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ε, για τον ΠΟΕ, με έναν άλλο εταίρο της Ανατολικής Ευρώπης στην Ουκρανία. Καθίσταται σαφές ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ε, ε, μεταξύ των αποτελεσμάτων. Πώς γίνεται ε, με την Ουκρανία να ήταν δυνατό να πείσουμε τον εταίρο μας ε, να περιορίσει κατά 50% τους εισαγωγικούς δασμούς, ενώ με τη Ρωσία συμφωνήσαμε να περιοριστούν οι δασμοί αυτοί εισαγωγών κατά μόλις 5%. έγιναν κάποιες ε, συμφωνίες εμπορικές με την Ουκρανία ε, λάβαμε κάποια ανταλλάγματα έλαβαν κάποια ανταλλάγματα ε, που δεν έλαβε η Ρωσία Επίσης, άλλε ερωτήσει που προκύπτουν είναι πώς γίνεται η Ρωσία να κατάφερε να διαφυλάξει αυτό το TRIMS για 7 ακόμη χρόνια με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις προμήθειες της εγχώριας αγοράς της τι προβλέπετε για το μέλλον των εμπορικών σχέσεων όσον αφορά τα μηχανοκινητά οχήματα. Μήπως είναι παράδοξο να προβλέπουμε τεράστια κέρδη για αυτό το τομέα της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ προετοιμαζόμαστε για ουσιαστικά μείωση των εξαγωγών ε, μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. Το τέταρτη ερώτηση είναι τα εξαρτήματα των ευρωπαϊκών οχημάτων ε, έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα εξαρτήματα. Θα βρίσκονται σε θεμητό ανταγωνισμό με όλες τις ε, χώρες που έχουν προσυπογράψει το επενδυτικό πρόγραμμα της Ρωσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αφού τίθενται ερωτήσει προ την Κομισιόν, θα επανέλθω σε εσά αργότερα για να απαντήσετε σε αυτέ τι παρατηρήσει και ερωτήσει. Α περάσουμε στον επόμενο εισηγητή. Τζαν Λούκα Σούστα από το SND, από του Σοσιαλιστέ, για την ε, συμφωνία στι συναλλαγέ στον τομέα των υπηρεσιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη εξήγησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα καθοριστεί μετά από την είσοδο της Ρωσίας, η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Το πλαίσιο αυτών των διμερών συμφωνιών είναι η ουσιαστική διατήρηση ορισμένων πλέον εκτιμάτων ε, ορισμένων ωφελών ε, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα χρόνια σε σχέση με ορισμένα ζητήματα. Το ζήτημα με το οποίο ασχολούμαι εγώ, όπως ε, αναφέρατε, σχετίζεται με τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τις προσωρινές μετακινήσεις ατόμων για, για επαγγελματικούς λόγους. Για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε αυτές τις ε, ε, συνθήκες, ε, τις πλεονεκτικές συνθήκες ε, όσον αφορά την εισαγωγή υπηρεσιών και το ίδιο μονογράφηκε αυτή η διμερής συμφωνία για τη διατήρηση ορισμένων αποκλειστικών πλεονεκτημάτων που είχε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 90 ώστε να αποφευχθεί ε, να υπάρξει περιορισμός αυτών των κανόνων μετά από την ένταξη στον ΠΟΕ. Ειδικότερα στην παρούσα περίπτωση αναφερόμαστε εκτός από τις θαλάσσιες μεταφορές σε 18 κατηγορίες επαγγελματικών υπηρεσιών. Η συμφωνία καθορίζει επίσης συνθήκες, προϋποθέσεις, αιτήσεις ποσοστώσεις ε, για την εργασία όπως αυτές έχουν δεσμευτεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συνεπάγεται νέα δέσμευση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά απλά επικύρωση της διατήρησης αυτής της πλεονεκτικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Ρωσία και η ε, Ρωσία δεσμεύεται ε, να ε, λάβει υπόψη στη ρήτρα της πλέον δεσπόζουσας χώρας. Ευχαριστούμε Τζαν Λούκα. Ο επόμενος εισηγητής είναι ο Ινέζε Βαϊντέρε για τις επόμενες δύο συμφωνίες για τους εξαγωγικούς δασμούς επί των πρώτων υλών και για τις εξαγωγές ξυλίας. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μιλήσω και για τις δύο εκθέσεις μαζί ή πρώτα για τη μία, πρώτα για την άλλη. Ε, θα προτιμούσα να ασχοληθώ ναι και με τις δύο ταυτόχρονα, αλλά μία-μία πρώτα, την πρώτη και μετά τη δεύτερη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε από κοινού με τις δύο αυτές εκθέσεις. Και η Ρωσία πρέπει να πάψει τις προστατευτικές ε, πρακτικές ε, που είναι κάπως συγκεκαλυμμένες βέβαια με το πρόσχημα της κρίσης και ούτω καθεξής. Και σε σχέση και με τη σχέση με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία. Για το πρώτο θέμα που είναι πρώτες ύλες, ε, για την ένταξή τη, στον ΠΟΕ δέχτηκε η Ρωσία να μειώσει ή να καταργήσει τους αγωγικούς δασμούς για κάποιες πρώτες ύλε. Τις δεσμεύσεις αυτές ε, τις ε, ολοκλήρωσε στο προηγούμενο πρόγραμμα παραχωρήσεων ε, προϊόντων, αλλά υπάρχει ένα κανθόδες θέμα. Με αυτόν τον κατάλογο δεν νομίζει η να καταργησει τους αγωγικου δασμου για καποιες πρωτες υλε τι δεσμευσει αυτες τι ολοκληρωσε στο προηγουμενο προγραμμα παραχωρησεων προιοντων αλλα υπαρχει ενα κανθοδες μπορεί να μην εισπράττει δασμούς για άλλα πρώτα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, σε αυτόν τον ε, κατάλογο. Η ρωσική κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην επανεισαγάγει ή αυξήσει εισαγωγικού δασμούς για έναν κατάλογο πρώτων υλών που θα περιλαμβάνει τις πρώτες ύλε που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πίνακα ε, των προϊόντων που συνήψε για να ενταχθεί στον ε, ΠΟΕ. και ιδίω ό,τι αφορά πρώτε που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οποίες υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό, σπόροι, γεωργικά προϊόντα, καπνών χημικές ουσίες, ε, μεταλλεύματα κτλ. κτλ. Δεύτερον, εάν εξακολουθεί να επιθυμεί να εφαρμόσει εξαγωγικού δασμού για αυτά τα προϊόντα, η Ρωσία θα πρέπει να έχετε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνε εκ των προτέρων για να λαμβάνει υπόψη ε, τι απόψει τη Κομισιόν, ώστε οι διάφορε συναλλαγέ να είναι προ όφελο αμοιβαίο. Δεν απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση. Το πρώτο μείζον πρόβλημα το οποίο εγώ βλέπω με το κείμενο αυτό είναι ότι δεν περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικούς περιορισμούς για την Ρωσία. Ε, το να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ιδίως έχοντας υπόψη τις εμπειρίες μας με τη χώρα αυτή. Επίση, δεν απαγορεύει σαφώ την υιοθέτηση νέων μέσων προστατευτικών από τη Ρωσία. Απλά λέει ότι θα πρέπει να έχει κάποια διαφύλαξη με την Κομισιόν εκ των προτέρων. Αλλά διαφωνήσει με οποιαδήποτε από τις ε, απόψεις της Κομισιόν, τι θα γίνει. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα και στις διαπραγματεύσεις για την νέα συμφωνία που θα αντικαταστήσει την PCA. Λέει η Ρωσία ότι έχει ήδη πληρώσει για την ένταξή της στον ΠΟΕ παρότι έχει συμφωνήσει όμως ευνοϊκούς όρους και μεταβατικές περιόδους. Επίσης δεν περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός ε, επίλυσης διαφορών σε αυτή τη συμφωνία και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να θέσω στην Κομισιόν κάποια ερωτήματα. Με ακούτε? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πρώτα απ' όλα ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση στα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα τα οποία ανέκριναν οι ρωσικές αρχές για το ζωικό κεφάλαιο, για τα ζώα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η απαγόρευση συνάδει με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα η εξέλιξη αυτή, η υιοθέτηση αυτών των μέτρων και δεν νομίζω ότι είναι συμβατά τα μέτρα αυτά με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ξέρετε ότι αυτό προκαλεί ανησυχία σε πάρα πολλού κτηνοτρόφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σε ό,τι αφορά τα, τις πρώτες Να έχουμε μία δεσμευτική για τη Ρωσία συμφωνία, ναι, αλλά πώς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον. Και αυτό είναι μια άλλη μου ερώτηση προς την Κομισιόν. Δεύτερη έκθεση τώρα, αν με επιτρέπετε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για τα προϊόντα ξυλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό που συνιστά μια σημαντική βελτίωση στην παροχή προϊόντων ξυλίας από την Ρωσία, η οποία έχει δεχθεί να μειώσει τους συντελεστές των εξαγωγικών της δασμών σε προϊόντα ξυλίας. Για κάποια είδη ξύλου έχει εισαγάγει κάποιες ε, δασμολογικές ποσοστώσεις εξαγωγές, χαμηλότερους δασμούς για την εξαγωγή και υψηλότερους ή από απαγορευτικούς δασμούς για όσα προϊόντα είναι πάνω από τις ποσοστώσεις. Ένα πρωτόκολλο μεταξύ Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο, στο παράρτημα της συμφωνίας αναφέρεται περί ε, κοινή διαχείρισης ε, των δεσμολογικών ποσοστώσεων. Υπάρχουν εφαρμοστικέ πράξει που έχει εγκρίνει η Κομισιόν. Η Ρωσία θα πρέπει λοιπόν βάσει αυτό να εκδίδει άδειε εξαγωγή ε, βάσει των σχετικών εγγράφων ε, εισαγωγή που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το πρωτόκολλο περιλαμβάνεται και η διαδικασία επίλυση διαφορών. Νομίζω ότι θα πρέπει να δεχθούμε να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία, διότι είναι ευεργετική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δεσμολογικέ ποσοστό με μειωμένου εξαγωγικού δασμού είναι κάτι που θα τονώσει σημαντικά ε, και την ε, επιπλοποιία και την ε, βιομηχανία ξύλια εν γέννη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα βασικό ερώτημα βέβαια είναι πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη. διότι έχουμε αυτές τις εξαγωγικές ποσοστώσεις που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρχε ε, σχετική νομοθεσία, επομένως πρέπει να δούμε πώς θα τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε την τελευταία. απόψε μεταξύ Επιτροπής και εισηγητών. Ας ακούσουμε τώρα και τους σκιώδεις εισηγητές για τις τέσσερις αυτές συμφωνίες. Τι κάνει το λόγο. Ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγητής για τις δύο τελευταίες συμφωνίες για τις πρώτες ύλες και για το ξύλο. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι. Θα ήθελα απλώ να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που εξέφρασαν και οι συνάδελφοι ήδη. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξη πιστεύω στο πλαίσιο του ΠΟΕ και ελπίζω, εύχομαι, η Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει το όντι της δεσμεύσης της, να συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της και κυρίως αυτές που απορρέουν από την ε, συμμετοχή της στον ΠΟΕ και ελπίζω να κρυθούν οι δύο συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ο πρόεδρος δεν ακούγεται. Η κυρία Βάντερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θέλω να επανέλθω ω σκιώδη τώρα εκ μέρου του ΕΛΚ ε, στο θέμα του εμπορίου στι υπηρεσίε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να υπογραμμίζουμε για την διμερή αυτή συμφωνία. Επιτρέπει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει προτιμησιακέ ε, σχέσει ε, παραχωρήσει εκεί που έχει ήδη προσδιορίσει τέτοιες σχέσεις όπως με τη Ρωσία από την ε, συμφωνία του 1994. Ε, Τι είδους προτεραιότητες όμως έχουμε ως προς την διαπραγμάτευση αυτών των ε, συμφωνιών, αυτής της συμφωνίας για τις υπηρεσίες και σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε στο 3 στις επενδύσεις επικοδομητική αντιμετώπιση του θέματος από τους Ρώσους, γιατί αυτό σημαίνει και για τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για τις τηλεπικοινωνίες και για πολλούς άλλους τομείς σημαντικές αλλαγές εκ μέρους της Ρωσίας προποθέτει δηλαδή μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες ενέργειας σε παραδείγματι που δεν είναι χωριστή ε, κατηγορία μέσα στις, στις γενικές συμφωνίες και που έχουν κοπεί σε διαφορετικές γραμμές που κατανέμονται σε άλλες υπηρεσίες επιχειρηματικών σχέσεων. Επί παραδείγματι, για την εξωτερική βιομηχανία ή για την διανομή. Σε διάφορου τομεί λοιπόν έχει κατακαιρματιστεί η ενέργεια. Ερωτώ τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια η Ρωσία ούτε στα οριζόντια ζητήματα ούτε και στι υποκατηγορίε των υπηρεσιών των σχετικών με την ενέργεια. Και το επόμενο ερώτημα είναι αν η νέα συμφωνία μπορεί να αποτελέσει δίωδο για μια επιτυχή και φιλόδοξη διατύπωση ε, προτάσεων συμφωνίας για την ενέργεια αργότερα. Έστω και αν δεν έχει προχωρήσει νομοθεσία σε παιδορωσικό. Πόσο μπορεί η Επιτροπή να πιέσει για το διμερές ε, εμπόριο. Φαντάζεστε βέβαια τι είδου αξία έχουν οι υπηρεσίε ενέργεια στη Ρωσία με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων και ε, όλων των υπηρεσιών της διανομής της εξωτερικής βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Λέω, Πρόεδρος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε παρά μόνο να πούμε ένα ναι ή όχι στις συμφωνίες αυτές, πρόκειται συμφωνίε συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και άρα μόνο να τις δεχθούμε ή να τις απορρίψουμε μπορούμε. Ερωτήσεις δηλαδή ή σχόλια δεν έχει πολύ νόημα να κάνουμε, εκτός και αν αποφασίσουμε εν τέλει να απορρίψουμε τις προτάσεις. Εάν κανείς άλλος συνάδελφος δεν θέλει ε, παρατήρηση, παρατηρήσεις ε, ή σχόλια. Πολύ ευχαριστώ στο λόγο τώρα στην Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις πρώτες παρατηρήσεις του κυρίου Ζαλεύσκη για το ζήτημα των κινητήρων και την προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα πολύ καλά για ποιο λόγο ανέφερε ότι με τη Ρωσία πετύχαμε μόνο μείωση 5% του δασμού διότι για τους εισαγωγικούς δασμούς αυτοκινήτων επιτύχαμε μείωση από 30% σε 15%. ή μάλλον είτε 50% ε, των δασμών, όχι όμως σε καμία περίπτωση 5%. Πρέπει να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή δεν, έχουν ακόμα, δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί μείωση των εξαγωγών ε, ευρωπαϊκών εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Ρωσία. Ίσα ίσα που τα στοιχεία που έχουμε ε, για το πρώτο τρίμηνο δείχνουν αύξηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Βάιντελε για τις ερωτήσεις της. Θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ακούμε πλήρως, αλλά μερικές φορές πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε ερωτήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Κατά πόσο υπάρχει η τάση προστατευτισμού στη Ρωσία και κατά πόσο βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση η κατάσταση με τη Λευκορωσία και το Βαζακστάν και κατά πόσο μας ενισχύει, ναι, η απάντηση είναι ναι. Τι κάνουμε για όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια νέα ακριβώς συμφωνία μέτρα πρόληψης ε, αυτή τη τάσης. Όσον αφορά ειδικότερα τι πρώτε ύλε, ο εισηγητή έχει δίκιο ε, όταν λέει ότι οι δεσμεύσεις της Ρωσίας δεν είναι νομικά δεσμευτικές και ότι απλά είναι δεσμεύσεις διαβούλευσης. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνω πόσο σημαντικές είναι οι νομικά δεσμευτικές ε, δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία για την ένταξή της για μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύψης της για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικοί εξαγωγικοί δασμοί έχουν, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό για τις μη υποχρεωτικές δεσμεύσεις ε, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις τουλάχιστον δύο μήνες ε, πριν. Όσον αφορά την ανησυχία για τη διαχείριση των ποσοστώσεων για την ξυλία, χτυπάμε ξύλο προς το παρόν. Τα πράγματα πάνε καλά και έχουμε ήδη μία ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής για την Ξυλία στις 23 Απριλίου. Μέχρι στιγμής ε, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Τέλος, ο εισηγητής μας ρώτησε επίσης κατά πόσο θεωρούμε την ενέργεια και τις υπηρεσίες ε, ενέργειας ε, σημαντικές. Ναι, φυσικά γνωρίζετε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων νέα συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι το κεφάλαιο της ενέργειας είναι μακράν το πιο δύσκολο κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, η οποία προς το παρόν αρνείται να ξεκινήσει μάλιστα τις συζητήσεις. Σαφώς, λοιπόν ε, είναι ένα από τα κέρια σημεία των συζητήσεων προς το παρόν ε, Πρέπει να γνωρίζετε ότι το έχουμε συμπεριλάβει ω αναπόσπαστο κομμάτι τη ατζέντα μα και δεν πρόκειται να τον καταλήψουμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ε, κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν δεν απάντησε στη σημαντικότερη ερώτησή μου για το ζωικό κεφάλαιο. Ε, άκουσα ένα παράπονο από τον Παύλ Ζαλεύσκη. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο, αν δεν έχετε πρόβλημα. Και μετά μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας, ώστε η Κομισιόν να επανέλθει σε αυτό, Παύλ Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή στρατηγική το να μην καταλαβαίνετε τις ερωτήσεις ε, όταν οι ερωτήσει είναι πολύ δύσκολε. Λοιπόν, θα την επαναλάβω, ώστε να, ε, να την καταλάβετε καλύτερα. Είπα ότι στην περίπτωση, στην περίπτωση της Ουκρανίας και ε, έδωσα συγχαρητήρια στην Κομισιόν για αυτό, η Κομισιόν κατάφερε στη συμφωνία με την Ουκρανία, να πει στην Ουκρανία να μειώσει του εισαγωγικού δασμού κατά 50%. Ε, Ξεκινώντα από ένα 10% το 2008 και προοδευτικά μειώνοντα αυτό το ποσοστό, ώστε το 2013, του χρόνου δηλαδή, να φτάσει στο τελικό επίπεδο του 5%. Αυτό ήταν δυνατό. Γιατί αυτό δεν ήταν δυνατό με τη Ρωσία. Τι μα έδωσε η Ρωσία ώστε να συμφωνήσουμε μαζί του κάτι εντελώ διαφορετικό. Και η συμφωνία αυτή είχε ω εξή. Η Ρωσία συμφώνησε να μειώσει του ε, εισαγωγικού δασμού κατά 5% έω το επίπεδο του 25% και θα διατηρήσει το 25% έως το 2018. Στη συνέχεια, μετά το 2018, το επίπεδο των δασμών θα είναι 15%. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τι κερδίσαμε από τη μία ανατολικοευρωπαϊκή χώρα και τι κερδίσαμε από τη Ρωσία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε λάβει κάποιο πολύ σημαντικό αντάλλαγμα σε κάποιον άλλο τομέα. Το η ερώτησή μου είναι τι κερδίσαμε σε έναν άλλο τομέα ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε μια τέτοια λύση η οποία ε, σίγουρα δεν είναι επωφελής ε, για τους παραγωγούς εξαρτημάτων μηχανοκινητών οχημάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Βάιντερε, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, έχω την εντύπωση μερικές φορές ότι η Επιτροπή συνεχίζει έναντι του στρατηγικού εταίρου να συμπεριφέρεται με φόβο μάλλον σοφοδέος και όχι σαν εταίρος ισότιμος. Αυτό το είπε και ο συνάδελφος μόλις τώρα και δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ έχω καταθέσει ερώτηση για το ζωικό κεφάλαιο και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνω απάντηση. Τα πρόσφατα λοιπόν περιοριστικά μέτρα που υιοθέτησαν οι ρωσικές αρχές για το ζωικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς τα βλέπει η Επιτροπή και είναι συμβατά με τις νέες δεσμεύσεις Ρωσίας μέσα στον ΠΑΕ. Επιτροπή είστε υπο... Είστε... Ε, δέχεστε επιθέσεις, μπορείτε να υπερασπιστείτε τους εαυτούς σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Ελεύσκη επεσήμανε τις σχέσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά δεν είναι ίδια εταίρε και δεν έγιναν συμφωνίες την ίδια χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν αχλάδια με μήλα, διότι οι εταιρικέ σχέσεις δεν είναι εν προκειμένου συγκρίσιμες μεταξύ των δύο αυτών κρατών. Με την Ουκρανία έχουμε ναι μείωση από το 10% στο 5%, με τη Ρωσία από 30% στο 15% των δασμών. Αλλά πάλι πρέπει να κοιτάξουμε το κάθε συγκεκριμένο προϊόν. Στα ελαφρά εμπορικά ε, οχήματα έχουμε, ιδιωτικής χρήσης, έχουμε από 25% στο 10% και για τα λεωφορεία το ίδιο έχουμε σημαντική μείωση. Αλλά, εάν θέλετε να συγκρίνετε τις δύο συμφωνίες μεταξύ τους, θα αποδείτε διαφορές από το ένα τομέα στον άλλο ασφαλώς. Πάντως, που σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ επωφελής για την ευρωπαϊκή οικονομία η συμφωνία αυτή με τη Ρωσία. Η δε συνολική μείωση δασμών σε ύψος αρκετών δισεκατομμυρίων είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτήν που μας προσφέρει συμφωνία με την Ουκρανία. Για την κυρία Βαντέρε δεν ε, ήθελα να αγνοήσω την ερώτηση σας, απλώς δεν πρόλαβα μέσα στο λίγο χρόνο που είχαμε στη θέσή μας. Έχουμε ήδη επισημάνει στις ρωσικές αρχές ότι η απαγόρευση εισαγωγών λόγω του πυρετού των χείρων ε, ήταν αδικαιολόγητη και παράνομη από άποψη του ΠΟΕ, μένα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει ότι δεν είναι ακόμη μέλος του ΠΟΕ η Ρωσία Το επισημαίνουμε μένα, αλλά σε διοικητικό επίπεδο. Δεν συμφωνούμε, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε και δεν δεχόμαστε αυτή την παράνομη απαγόρευση εισαγωγών. Ευχαριστώ, λίγο πρόεδρο. Σας ακούσουμε ίσως κάποια σύντομα σχόλια από τους οι εισηγητέ. Πρέπει να σας πω επίσης ότι έχουμε μια ομάδα παρακολούθησης των σχέσεων με την Ρωσία στη υπό τον εισηγητή κύριο Ρόμπερτ Στέρντι και αποφάσισαν χθε οι συντονιστέ στην ημερήσια μας διάταξη να συμπεριλάβουν και την παρακολούθηση των διαδικασιών για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Και βεβαίως μπορούμε να ε, συντάξουμε και να εγκρίνουμε ψήφισμα στο θέμα αυτό. Ο κύριο Ζολεύσκη έχει το λόγο για να ξαναρχίσουμε με τους Θα μιλήσω αγγλικά για να είμαι πιο ξεκάθαρη. Δεν ήταν ε, μείωση το 10% αυτή για την Ουκρανία. Από το 25% πήγε στο 10% και τώρα είναι γύρω στο 5%. Αυτό ήθελα να πω. Σας ζήτησα ποια είναι τα δυνητικά κέρδη που έχουμε εμείς αποκομίσει άλλους μέσα από τη Ρωσία. Δεν θέλω Κι εγώ σε καμία περίπτωση να συγκρίνουμε τα μήλα με τα χλάδια, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Η δική μου πρόταση είναι η εξή. Ξεκινά μια νέα εποχή στις εμπορικές μας σχέσεις με τη Ρωσία. Όταν δηλαδή θα γίνει μέλος του ΠΟΕ η Ρωσία. Η πρότασή μου λοιπόν είναι θα ήταν συνετό να συντάξουμε ένα γενικό ψήφισμα για τις εμπορικές μας σχέσεις με τη Ρωσία στην νέα αυτή κατάσταση, να συζητήσουμε στην Ολομέλεια και να συμπεριλάβουμε στο ψήφισμα τις παρατηρήσεις τις οποίες είχαμε διατυπώσει και στην προηγούμενη συζήτηση, όπως και σε αυτή, ε, για μια σειρά ιδιαίτερα λεπτών ζητημάτων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε το ενδεχόμενο συντάξης ενός γενικότερου ψηφίσματος για τις εμπορικές μα σχέσεις με τη Ρωσία. Να μην επικεντρωθούμε δηλαδή μόνο στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία συζητήσαμε και σήμερα αλλά και πρόσφατα. Ευχαριστώ. Τζον Λούκα Σούστα, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Όχι. Δεν έχετε κάποια άλλη. Κύρια Βάιντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα να πω ε, δεν είναι αν θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι, μάλλον ναι πρέπει να πούμε. Πάντως οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές απόψε είναι πολύτιμες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ζαλεύσκη να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάρτιση ενό ξεχωριστού ψηφίσματος για τις εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία, όπου να μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψει μας. Αυτή την απάντηση σα αν είμαστε στην Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρο. Ωραία, να Ας περάσουμε στο σημείο 17. Ε, αυτό το είναι ένας κανονισμός για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ονομάζεται κανονισμός ICI. Αποτελεί απάντηση στον κανονισμό ICI που αυτή τη στιγμή αποτελεί το κύριο μέσο για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανεπτυγμένες χώρες. Ο εισηγητής μας... Ε, είναι ο Λάιμα Λιουσία Αντρικένε από το ΕΛΚΑ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά έχουμε μόνο 7-8 λεπτά πριν από την ψηφοφορία. Μπορώ να σας ζητήσω να συζητήσουμε αυτό το σημείο μετά από την ψηφοφορία, διότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Δυστυχώς είναι υπερφορτωμένο σήμερα η ημερήσια διάταξη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με το ε, σημείο αυτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή μας ε, πρέπει να παρουσιάσει, ζητήθηκε από την Επιτροπή μας να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση. Παρακαλώ κάντε ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. ζητήθηκε από την Επιτροπή μας να παρουσιάσει μια νομοθετική έκθεση για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δημιουργεί ένα μηχανισμό εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες. Η κυρία πρόκληση που αντιμετωπίζει ο προτινόμενος μηχανισμός αποτελεί συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. Το πλαίσιο της παγκοσμίας οικονομίας έχει αλλάξει, οι εξουσίες έχουν αλλάξει, η ευημερία διαδίδεται όλο και περισσότερο και δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον στο διεθνές προσκυνείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν είχε αυτή τη στιγμή μηχανισμό με τον οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες αναδυόμενες δυνάμεις σε ζητήματα που σχετίζονται ε, με την πρόθεση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντιμετώπιση ε, παγκόσμιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή αυτή η συνεργασία είναι δυνατή στο πλαίσιο του μηχανισμού ICI ε, που ωστόσο περιορίζεται σε 17 υψηλά βιομηχανοποιημένες χώρες ή χώρες ε, υψηλών εισοδημάτων όπως είπα Κορέ, ε, Νότια Κορέα η συνεργασία με χώρες όπως Κίνα, Ινδία και Βραζιλία εντάσσεται στο μηχανισμό συνεργασίας για την ανάπτυξη σημαίνει ότι αυτό η συνεργασία περιορίζεται σε δράσεις που σχετίζονται με την ε, εξάλληψη της φτώχειας ε, στις ε, δικαιούχους χώρες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο μηχανισμό για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Το πρωτενόμενος μηχανισμός συνεργασίας που αποτελεί κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ μιλάμε για οικονομική υπάρχει ε, οικονομικό πλαίσιο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ε, ευρώ από το 2014 στο το 2020. Αυτός ο κανονισμός θα αντικαταστήσει το χρηματοδοτικό μέσο συνεργασίας για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, το ICI-SA+, που λυγεί το 2013. Ωστόσο, το Μηχανισμό Συνεργασία για την Ανάπτυξη και το Μηχανισμό Ευρωπαϊκή Γειτονία και Προενταξιακή Βοήθεια θα συνεχίσουν και στο διάστημα 2014-2020. Ο μηχανισμός συνεργασίας θα πρέπει να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει στόχους πέραν απλά της συνεργασίας για την ανάπτυξη για την πρόθεση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού στον κόσμο και για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων όπου απαιτείται. Έχει λοιπόν ο μηχανισμός τρει κύριου στόχους. Πρώτον, η υλοποίηση της διεθνούς διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μέχρι της υποστήριξη των διαφόρων στρατηγικών συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, βελτίωση τη πρόσβαση στην αγορά και ανάπτυξη του εμπορίου και των ευκαιριών εμπορικών συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τρίτον βελτίωση της κατανόησης ε, ε, των μειονεκτημάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόθεση των συνεργασιών. Όλα αυτά για την υποστήριξη ε, πολιτικών όπως της εμπορικής πολιτικής και της εξωτερικής διάστασης, της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης των κοινωνικών πολιτικών καθώς και των ε, τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Την περασμένη εβδομάδα είχα μια πρώτη συνάντηση με την ε, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για τα μέσα εξωτερικής πολιτικής και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης διατύπωσα την υποστήριξή μου για την ανάγκη αυτού του νέου μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής αλλά εξέφρασα και τους μεγάλες μου ανησυχίες που θα ήθελα να επαναλάβω εδώ σήμερα. Η κυρία μου ανησυχία είναι ότι αυτό το ο μηχανισμός δεν θέλω να είναι πολύ, να εντάσσεται πολύ σωστά μεταξύ των υπολείπων μηχανισμών και να συντονίζετε σωστά με αυτούς. Δεύτερον, έχει τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων σε πολλές περιοχές αλλά περιορισμένο προϋπολογισμό. Το άρθρο 2 μιλάει για το πεδίο εφαρμογής που σύμφωνα με το κείμενο είναι όλες οι τρίτες χώρες, περιφέρειες και εδάφη. Όλες οι τρίτες χώρες, οι περιφέρειες και τα εδάφη μπορεί να είναι επιλέξιμα. στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι υποστηρίζονται μέτρα συνεργασίας με αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες όπου έχει ιδιαίτερα συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι με τον ετήσιο προπολογισμό 160 εκατομμύριων ευρώ θα πρέπει να στοχευτούν πολύ σωστά οι περιφέρειες και τα εδάφη. Αυτό που με ανησυχεί λοιπόν είναι πώς οι στόχοι, οι προτεραιότητες, οι περιφέρειες, οι χώρες και τα κονδύλια πρόκειται να προσδιοριστούν. Ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι τα γεωγραφικά και τα θεματικά προγράμματα στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού και ποιες είναι οι χώρες ε, μπορούμε ήδη να αναφέρουμε στο κείμενο του κανονισμού τις χώρες οι οποίες ε, έχουν σχέση με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, δεν βρήκα μέσα στο κείμενο διατάξεις για τη διαδικασία επιφύλαξης εξέτασης όσον αφορά το πολιετές ε, πρόγραμμα και τους στόχους και τα κονδύλια. Αναφέρεται σε ένα άλλο όρθρο ότι πρέπει να καθορίζεται καθαρά μια στρατηγική για μια συγκεκριμένη χώρα ή για μια περιφέρεια. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μηχανισμού συνεργασίας αναφέρεται ότι έχει, θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο έγγραφο για κάποιες χώρες και έτσι τα ο πολιτή προγραμματισμό θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό το έγγραφο. Θέλουμε η Κομισιό να μας εξηγήσει σε ποια νομική βάση και πώς συντάσσεται αυτό το κοινό έγγραφο και πώς θα εξετάζεται το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού. Τέλος, στο άρθρο 5, παράγραφος 6, όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης, γίνεται αναφορά σε μη ουσιαστικές τροποποιήσεις των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων. Ε, μια διαδικασία εξέτασης δεν θεωρείται διαδικασία εξέτασης όταν αυξάνει ή μειώνει κατά περισσότερο από 20% το συγκεκριμένο κονδύλιο. Θα ήθελα να μας εξηγήσει αυτή, η Κομισιόν πώς ε, καθορίζεται αυτό το 20%. Επίσης ήθελα να τονίσω ότι ο συνολικός προπολογισμό αυτού του μέσου είναι 1,13 δις ευρώ. Θα είναι ωστόσο λιγότερο, διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 η χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus for All εντάσσεται σε αυτόν τον κανονισμό. Επίσης θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσει η Κομισιόν πώς θα ενταχθεί το Εράσμους ε, και τι ποσοστό του προπολογισμού αυτού του μέσου θα κατανεμηθεί, θα εκχωρηθεί στο Εράσμους. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό έγγραφο, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι θα πρέπει να φροντίσουμε να χρησιμοποιηθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται ο προπολογισμό. Πριν καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτή την πρόταση, θα πρέπει να έχουμε μια σαφή απάντηση ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του ε, μέσου και πώ θα επιτευχθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέσατε πολλά ερωτήματα προς την Κομισιόν. Είμαι βέβαιος ότι τα έχετε, κύριε πρόσωπο της Κομισιόν, σημειώσει. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σούστα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συντομία, διότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κάνω μια πολιτική ερώτηση. Πιστεύω ότι και σε αυτό το θέμα θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα με άλλες ε, επιτροπές όπως με την ΑΦΕΤ ε, περί αρμοδιότητας. Όλες οι επιτροπές εδώ και όλες οι ομάδες του Κοινοβουλίου και όλοι οι πρόεδροι θα υπερασπίσουν αυτή την, ε, το θέμα της αρμοδιότητας. Το δεύτερο θέμα εμείς γνωρίζουμε ότι όλα τα, όλοι οι μηχανισμοί συνεργασίας, βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις τρίτες χώρες, είναι θεμελιώδης σημασία για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο όσον αφορά την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία κανόνων ελεύθερου εμπορίου, θεμητών κανόνων και τη προστασία των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και για την ενίσχυση τη διμερούς συνεργασία σε στρατηγικού τομεί ε, στους οποίου εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δέσμη μέτρων αφορά κονδύλε 70 δισεκατομμυρίων για... Ε, ο μηχανισμός για τον οποίο μιλάμε τώρα είναι πολύ μικρός αν μιλάμε για μόλις ένα δις αρκετά μειωμένος προπολογισμό σε σχέση με τους στόχους που τίθενται. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο μηχανισμός αποτελεί διάδοχο του ICI και είναι ανοιχτός σε όλες τις τρίτες χώρες, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει επίσης βάσει των δικών της κοινοτικών συμφερόντων ποιες θα είναι οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα εκχωρηθούν οι πόροι, ποιοι τομείς πρέπει να ληφθούν υπόψη και ποιοι επίσης είναι οι τύποι επιχειρήσεων προς τους οποίους θα προσανατολίσουμε κυρίως ε, τις ενισχύσεις μας. Και εκεί έχουμε μια τελευταία πολιτική σκέψη. Εμείς ε, είδαμε εκεί που συζητήθηκε το ICI να γίνεται ένα brand fair μεταξύ της ε, Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για τις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε οι ορισμοί αυτών των νέων εργαλείων, νέων μέσων να μην περιορίζονται μόνο στο να αποτελούν ένδειξη δύναμης, αλλά να ε, βοηθούν επίσης ε, στη δημιουργία προϋποθέσεων με τις στις ανταλλαγές με τις τρίτες χώρες ε, που θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο στο πλαίσιο της υπάρχουσας δομής του υπάρχοντος μηχανισμού να καθορίσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Δηλαδή αυτή τη συμφωνία που πετύχαμε πριν από μερικούς μήνες για το ICI Plus και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα και να φροντίσουμε να μην αναπαραχθούν οι αρνητικές πτυχές που είχαν εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα την Κομισιόν. Υπήρξαν ε, ενστάσεις, ερωτήματα που έθεσε κύριος η Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γκάρι Μίλλερ από την Κομισιόν. Ησυχία παρακαλώ. Thank you. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Not showing the respect that we should pay. Παρακαλώ δεν δείχνουμε τον δέοντα σεβασμό προς ομιλητές και και σας παρακαλώ να καθίσετε αγαπητοί συνάδελφοι και μην ε, συζητάτε μεταξύ σας. Παρακαλώ να ακούσετε τους ομιλητές. Δείξτε το δέοντα σεβασμό. Παρακαλώ. Starting with some respect for the chair. Δείξτε πρώτα σεβασμό στον πρόεδρο και μετά και στους ομιλητές. Παρακαλώ, κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιτέλους συζητάμε αυτή την πολύ σημαντική πρόταση στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Καταρχάς να μιλήσω εν συντομία για το ποιο κάνει τι. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως είπε και η κυρία Αντρική, έχουμε την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η οποία ε, στενά συμμετείχε στην εκπόνηση της πρότασης ε, που συζητείται εδώ σήμερα. Πρόκειται όμως για πρόταση της Κομισιόν και όπως είπε και η κυρία Αντρικίν είμαι ε, είναι στην υπηρεσία για τις, ε, τα μέσα εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε υπό την αιγίδα της ΥΠΑ εκπροσώπου, κυρία Σάστον, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτήν την μονάδα όπως και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε συγκροτήσει λοιπόν μια ομάδα και είμαστε στην διάθεση της Επιτροπής σας ε, για να προχωρήσουμε από κοινού. Όπως είπε και η συγγήτρια, οι συνάδελφοί μου είχαν ήδη επαφές μαζί της και συζήτησαν την πρόταση. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να τονίσω ότι ο μηχανισμός εταιρικής σχέσης που προτείνουμε είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία και δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Εάν ε, δει κανεί ε, τα άλλα μέσα, τους άλλους μηχανισμούς του όλου πακέτου, ε, λίγο πολύ είναι όμοια με αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής. Με αυτό, το μηχανισμό, με αυτό το νέο μηχανισμό εταιρική σχέση θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα μέσο, ως ένας μηχανισμός και αυτό πιστεύω ότι μεταφράζει στην πράξη τις προσδοκίες που γεννούνται μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας και εντάσσεται στην εργαλειοθήκη της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι βουλευτές ανέφεραν το μέσο για τις ε, εκβιομηχανισμένες χώρες. Έχουμε αυτό το μέσο για αρκετές εκβιομηχανισμένες χώρες. Ε, το ICI Plus αναφέρθηκε και αυτό. Είναι ένα μηχανισμό που μα δίνει τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε αντίστοιχα project και σε αναπτυσσόμενε χώρε. Να τονίσω όμω για μια ακόμη φορά ότι με αυτό το μηχανισμό θέλουμε να προχωρήσουμε έτσι περαιτέρω και να μπορούμε να προωθήσουμε τα σφαίροντά μας σε παγκόσμιο επίπεδο ε, σε μια ευρία γκάμα θεμάτων και τομέων. Η συνάδελφο μου από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να σα δώσετε το λόγο, θα σα δώσουν κάποια παραπάνω στοιχεία. Ποια είναι τα βασικά όμω ε, χαρακτηριστικά αυτού του νέου μηχανισμού και επειδή έγιναν και σχόλια ε, από συγκεκριμένους βουλευτές, να σας πω ότι ε, θέλουμε να έχει κάποια βιώσιμα στοιχεία, με βασικότερο την ευελιξία. Έχουμε λοιπόν την επταετή περίοδο αυτή, στη διάρκεια τη οποία θέλουμε να έχουμε ένα μηχανισμό που θα δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να δρά γρήγορα σε ένα ταχαίω ε, μεταβαλλόμενο διεθνέ περιβάλλον, αμεταλλασβολόμενε ανάγκε, αλλά αλλάζουν και οι εταίροι. Στη διάρκεια αυτή τη επταετία, οι στρατηγικέ μα σχέσει ενδέχεται να αλλάξουν να μεταβληθούν. Εξού και πιστεύουμε ότι χρειάζεται η ευελιξία στην υλοποίηση του μηχανισμού αυτού για να μπορέσουμε να αποκριθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιες προκλήσεις. Το θέμα ε, των μη ουσιοδών τροποποιήσεων ε, ακριβώς εδώ ε, πρέπει να συζητηθεί. Θέλουμε λοιπόν ευελιξία στην υλοποίηση του μηχανισμού και είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με την Επιτροπή σας για να σας εξηγήσουμε γιατί είναι αυτό απόλυτα απαραίτητο. Όπως είπε η συγγήτρια, θα εστιάσουμε στις αναπτυγμένες, αλλά θα έχουμε σχέσεις και με αναπτυσσόμενες χώρες. και γιατί έχουμε στρατηγικό ε, συμφέρον και ενδιαφέρον. Υπάρχουν αλλά και ε, κάποιε αναπτυσσόμενε χώρε που αναδύονται στο παγκόσμιο προσκήνιο και διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Ποιε θα είναι οι δράσει μα βασικά λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Δεν θα είναι κλασική αναπτυξιακή βοήθεια. δώσω το λόγο στον συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που υπόθηκε σε σχέση με τον προπολογισμό, αν επαρκεί δηλαδή. Δύο σχόλια και ολοκληρώνω με αυτά, κύριε Πρόεδρε. Πρώτο σχόλιο. Όταν δεν τυπώσαμε την πρόταση, κάναμε τους υπολογισμού, κάναμε μια μελέτη επιπτώσεων, αναλύσαμε λεπτομερέστατα τι νομίζουμε ότι θα χρειαστεί ε, σε αυτή την επταετία και φτάσαμε σε αυτό το νούμερο, το οποίο βέβαια θα συζητηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο όλων των μηχανισμών, κατηγορίο, στην κατηγορία 4, εξωτερικές δράσεις. Με αυτό το ποσό όμω το οποίο έχουμε ζητήσει, πιστεύουμε ότι θα έχουμε επαρκή πόρου στη διάθεσή μα, αλλά ευχαρίστω να τα συζητήσουμε. Και αν θέλετε να επιχειρηματολογήσουμε ευχαρίστω, μήπω και σα πείσουν. Πρέπει να καταλάβετε πάντως ποια είναι η φύση αυτού του μηχανισμού. Δεν είναι κλασικό ε, μηχανισμός αναπτυξιακής ε, συνεργασίας και βοήθειας. Δεν θα έχουμε δημιουργία θεσμών ε, και δημιουργία υποδομών σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ουσιαστικά οι δραστηριότητες θα διαφέρουν. Θα είναι μικρή κλίμακα, θα είναι ευέλικτε, εκφύσεως. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία τα οποία εγώ θα ήθελα να τονίσω θα δώσω όμως το λόγο στη συνάδελφα Φερνάντε από την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να συμπληρώσει αυτά που είπα εγώ. Αλλά όπως είπα, προσβλέπουμε στην συνεργασία μας με την δική σας επιτροπή και στο μέλλον. Μάλιστα. <clears throat> Ευχαριστώ κι εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστούμε που είμαστε στη θέση που μας επιτρέπετε σήμερα να παρουσιάσουμε αυτές τις προτάσεις στο Κοινοβούλιο. Είμαι επικεφαλής ε, του τμήματος ε, ε, η για τις προτάσεις, όπως ξέρετε, που έχουν σχέση και με τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Έτσι λοιπόν, όπως και με το σχεδιασμό μας, διατυπώνουμε κείμενο προτάσεων της ε, Επιτροπής εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δέχομαι βεβαίως ε, και κατανοώ τις του εισηγητού, είναι κοινέ σε όλους. Δεν θέλω να επισημάνω ότι αυτό το μέσον για πρώτη φορά προτείνει την προστασία και προαγωγή συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα έχουμε προσδιορίσει σε σχέση αμοιβιότητας με τους εταίρους και στρατηγικούς εταίρους και τις αναδυόμενες κοινωνίες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο πολιτικής, γιατί προσδιορίζεται, χαρακτηρίζεται και στη συνέχεια μπορεί να γίνει συζήτηση για τους τομείς της συνεργασίας, έχετε δει και εσείς, έχει εντοπίσει πιστεύω και ο εισηγητής, κάποιος από αυτών των οποίων ορισμένα έχουν μεγάλη σημασία για την Επιτροπή σας, του, ε, τα εμπορικά θέματα δηλαδή, αλλά όπως θα δείτε δεν πρόκειται μόνο για θέματα εμπορικά. Έχουμε να κάνουμε με ένα μέσο χάραξης πολιτικής που στόχο έχει να προαγάγει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε διάφορους τομείς πολιτικής, σε διάφορους τομείς συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τις θέσεις στον κόσμο και με τον οποίο προσπαθεί να προαγάγει τη θέση της στον κόσμο, είτε πρόκειται για την παγκόσμια οικονομία, τη γεωστρατηγική, τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή με τις κλιματικές αλλαγές. Έχει αλλάξει ο κόσμος, πολλές μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, μεγάλες χώρες οι οποίες διεκδικούν μερίδιο μερίδιο και πολιτικό, δηλαδή βούληση και ικανότητα, όπως λέμε σε εθνείς σχέσεις, για ανάληψη διπλωματικής δράσης, δράση στο διπλωματικό επίπεδο και αυτό βεβαίως αντιλαμβανόμαστε και ανταποκρινόμαστε σε αυτό το δεδομένο. 1,13 δίσσα, ε, ως ποσό, ίσως φαίνεται μάλλον ταπεινό σε σχέση με το μέγεθος του εγχειρήματος. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος μου τώρα, δεν χρειάζεται η ίδια χρηματοδότηση για υποδο... όπως με τις υποδομές ή την κοινωνική προστασία ή με την ε, διακυβέρνηση σε τρίτες χώρες, τον υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες αυτές, όπως όταν υποστηρίζουμε απλώς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ακούω τις παρατηρήσεις του εισηγητή και την ανησυχία του για διαφοροποίηση σχέση με άλλα μέσα. Θα ήθελα να πω ότι εδώ ιδιαίτερη, ιδιαίτερη σημασία έχει η προαγωγή των δικών μας ε, των ευρωπαϊκών ε, συμφερόντων εκτός OGA, ένα ICI Plus θα έλεγα, αλλά και πέραν αυτού θέλουμε να πλησιάσουμε και άλλες χώρες και κατά τρόπο στρατηγικό. Επομένως πρέπει να προσδιορίσουμε, να εντοπίσουμε ως στόχο των επιλογών αυτών συγκεκριμένες χώρες, αλλά και να διαρωτηθούμε εάν τα συμφέροντά μας θέλουμε να τα προωθήσουμε και σε άλλες χώρες ή περιοχές του κόσμου, έστω και αν δεν έχουν τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας ή στρατηγικής σημασίας. Ο εισηγητή νομίζω ότι ξεκάθαρα επισήμανε αυτό που είναι κοινό, πιστεύω, στο μυαλό όλων μα, ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, Κίνα, Ινδία, ε, Ιαπωνία. Πρέπει ωστόσο και να είμαστε σε θέση να προαγάγουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλε χώρες πέραν αυτών. Θα ήθελα και άλλα πράγματα να πω, αλλά νομίζω ότι έχει λήξει ο, χρόνος μου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς έχει στήσει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά την συγκεντρία. Είναι πολύ σημαντικό το μέσον αυτό που μας απασχολεί. Μια δουλειά στο ICI και ICI Plus τόσων ετών πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει με τον τριμερή διάλογο, Συμβούλιο και Επιτροπή δηλαδή για την περαιτέρω ανάπτυξη των σημαντικών μέσων. Και θα συνεχίσω στα λόγια του εκπροσώπου της πίεση Εξωτερικής Δράσης για να πω ότι όταν έχουμε μεγάλους στόχους, ευρύς στόχους, θα πρέπει ξεκάθαρα να λέμε ότι κάνουμε ισότιμα και την προσπάθεια για ένα αναπτυξιακό μέσον. Δηλαδή αναγνωρίζουμε και τα συμφέροντα των κρατών εκείνων που θέλουν να αναπτύξουν την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πριν από δύο-δυόμιση χρόνια είχε ξεκάθαρα πει ε, ότι αλλάζει στάση σε σχέση με το παρελθόν και είχε καταθέσει πρόταση στο Κοινοβούλιο με αρκετό χρονικό περιθώριο ώστε να ε, μελετήσουμε κι εμείς και να επεξεργαστούμε σε επίπεδο της δικής μας επιτροπή και γνώτερα του Κοινοβουλίου τις ε, προτάσει αυτές. Και θα ήθελα στον κύριο Σούστ να πω ότι είχε πολύ δίκιο ότι στο θέμα των της συνεργασίας δηλαδή με τις άλλες επιτροπές θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερνάντες ήταν ο πρόσωπος της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εξωτερικού Εμπορίου, Εξωτερικών ε, Σχέσεων. κύριε Αντρικένε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις που έδωσαν. Είμαι φυσικά έτοιμη να δεχτώ όλες αυτές τις εξηγήσεις, ε, να τις λάβω υπόψη μου κατά την εργασία αυτού του σχεδίου. Αυτός ο κανονισμός είναι καινοτόμος. Ε, διαφέρει από τα μέσα εξωτερικής δράσης. Καταλαβαίνω επίσης ότι το βασικό στοιχείο είναι η ευελιξία, αυτό που αναφέρθηκε. Μέσα στην αιτία, οι στρατηγικοί εταίροι μας μπορεί να αλλάξουν, γι' αυτό χρειάζεται ευελιξία. Ταυτόχρονα, κοιτάζοντας τα κονδύλια, το προϋπολογισμού στο ε, νέο δημοσιονομική προοπτική μιλώντας για αυτά τα μέσα που ανέφερα προηγουμένως ε, η εξωτερική διάσταση είναι 56 δισεκατομμύρια ευρώ η προενταξιακή βοήθεια 14 δις ε, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας 23 Υπάρχει μεγάλη διαφορά λοιπόν μεταξύ αυτών των κονδυλίων. Τα ερωτηματικά μου λοιπόν παραμένουν. Καθώς εδώ βρισκόμαστε σε πρωταρχική ανταλλαγή απόψεων, σε συνεργασία με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε συμβιβασμό. Ε, επόμενη εξέταση 23 Απριλίου. Ε, έχουμε τώρα ψηφοφορία. Έχουμε εκατοντάδες ε, θέματα για να αποφασίσουμε, για να ψηφίσουμε. Μια ανακοίνωση όσον αφορά την προθεσμία τροπολογιών. Χθε είδαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρατείνουμε την προθεσμία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση επειδή αυτό αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης και αποφάσισαν να παρατείνουν την προθεσμία. Μπορούμε λοιπόν να παρατείνουμε και εμείς τη δική μας προθεσμία. Τροπολογίες λοιπόν για αυτό το αρχείο μέχρι τις 23 Απριλίου 6 το απόγευμα. 6 μετά μεσημβρίας. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Προετοιμάστε τις κάρτες σας και προετοιμαστείτε και εσείς να ψηφίσετε. Το πρώτο αρχείο είναι μια γνωμοδότηση, το σημείο 18, ε, Ανάπτυξη συνεργασίας στην ενεργειακή πολιτική, εισηγητής Γιάννη Ζαγραντέλ. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Προφορική τροπολογία 1. Αντιρρήσεις. Στην προφορική τροπολογία καμία ψηφίζουμε Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήματική ψηφοφορία για την παράγραφο 5. Πρώτο κομμάτι, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι, ας ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πολύ εύκολη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση. Σχέδιο γνωμοδότησης για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους με τον κύριο Ιακολίνο. Συμβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμών 3. Υπέρ κατά αποχές. Ας ψηφίσουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεκατέσσερα, δεκατέσσερα υπέρ, κατά, αποχές δεν βλέπω πως ψηφίζουν οι φιλελεύθεροι, παρακαλώ να σας δω. Ε, υπέρ δηλαδή. Καλ... Εγκρίνεται τότε. Όχι να επαληθεύσουμε στην 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Οι φιλελεύθεροι λύνουν και δένουν, όπως ξέρετε. Ανεβάζουν και κατεβάζουν. Επομένως, προσοχή στην 3. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά καταπέπτει. Και πάμε στην 29. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απερίφθη. Η τροπολογία 29. Να επαληθεύσουμε την 29, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Αμάν, λέει ο πρόεδρο. Ξεκάθαρο το λάθος μου. Οι 30 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Επαληθεύουμε το δεύτερο κομμάτι παρακαλώ. Υπέρ. Ε, ψηφοφορία μάλλον. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Όχι, ε, γυρνάω στην 40 λέει ο πρόεδρος και την επαληθεύουμε. Αρχή ψηφοφορία, πέρασε ψηφοφορία. εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο σύνολο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίνεται 27 υπέρ. Μία ψήφος κατά δύο αποχές και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάω στο σημείο 20. Νομοθετικό θέμα, μάλλον δέσμη νομοθετική, Omnibus 2, με μεγάλη σημασία, γι' αυτό προσέχετε πώς ψηφίζετε. Συμβαστικές τροπολογίες 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Τρίτο μπλοκ τροπολογιών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τέσταρτη δέσμη υπέρ κατά εγκρίνεται. Μπλοκ παριθμών 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστικό μπλοκ, συμβαστική δέσμη 1 καταπίπτει. Συμβιβαστική δέσμη 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πώς μου αρέσει να περνάνε όλα αυτές τι σελίδες. Πάμε στη συμβιβαστική 4. Υπέρ. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Τέσσερα. Σας το δείχνω και με τα δάχτυλα. Υπέρ. Page 7. Είναι στη σελίδα 7 κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πιστεύεστε τον πρόεδρό σας. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέσμη 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στις αιτιολογικές σκέψεις στα recitals τροπολογία 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Α, όχι. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σχεδόν ομόφωνα εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ και μια αποχή. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και αυτή τη φορά ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Στην άλλη κάποιος ψηφίζει παραπάνω. Τώρα κλείνει η ψηφοφορία. Το ίδιο αποτέλεσμα, 28 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Συγχαίρουμε τον εισηγητή για τεράστια αυτή επιτυχία. have to vote. Λοιπόν, πρέπει να μας πει ο εισηγητής τώρα τι προτείνει. I have... Uh, uh, thank you very much, Mr. Κύριε Πρόεδρε, επειδή λίγο πολύ συμφωνήσαμε όλοι ότι θα μπορούσαμε πλέον να περάσουμε στις ανεπίσημες επαφές με το Συμβούλιο, αυτό θέλω να σας προτείνω να κάνουμε. Proposal πρόταση είναι λοιπόν να ξεκινήσουμε σαν επίσημες διαπραγματεύσεις ε, με το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν ε, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας στην πρώτη ανάγνωση. Βέβαια, η έκθεση όπως τροποποιήθηκε θα αποτελέσει τη βάση διαπραγμάτευσης της διαπραγματευτικής ομάδας. Που ήθιστε θα απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον εισηγητή κύριο Λάχτφριντ τους σκιώδεις εισηγητές Κοχμερίνα, Κρίστα Ρότβολ, Στέρντι, Σόλτς. Να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Let's move to the next Περνάμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Υπαρχόν 21. Legislative file. On uh, certain restrictions περιορισμοί για την εισαγωγή ορισμένων ε, πρώτων χάλιβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία, εισηγητή ο Ρόμπερτ Στέρντι. Ας ψηφίσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Άρα περνάμε απευθείας στην ψηφοφορία επί της πρότασης της Κομισιόν που δεν έχει καμία τροπολογία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα υπέρ. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Και πάλι ομόφωνα δεκτή η πρόταση δεν είναι και συνηθισμένο. Συγχαρητήρια κύριε Στέρτη και περνάμε τώρα στο όχι. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε. Έχω μία πρόταση λοιπόν από τον εισηγητή να έχουμε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για Συμφωνία σε Πρώτη Ανάγνωση. Η έκθεση που μόλις εγκρίναμε θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα διαπραγματευτεί η ομάδα μας, η διαπραγματευτική ομάδα. Αν καταλήξουμε σε συμφωνία, το σχέδιο έκθεσης θα κατατεθεί απευθείας στην Ολομέλη για να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση. Η διαπραγματευτική ομάδα θα απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον εισηγητή κύριο Στέρντι και τους Σκιώδης. Παύλ Ζαλεύσκη, Κούτας, Κοχμερίν, τη Τέιλορ, Σόλτς. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο Ντανιέλ Κάσπαρ θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Πολύ δυσάρεστο μου είναι να το ομολογήσω, αλλά στα δύο πρώτα σημεία, 18 και 19 των ψηφοφοριών, ε, είχαμε μόνο μία ψήφο διαφορά, στην, ε, με αποτέλεσμα την έγκριση τελικά για την απόρριψη. Ξέρετε όμως ότι έχουμε ένα μέλος με επιπλέον ένα μηχάνημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν δεχόταν την αρνητική ψήφο από ό,τι μας είπε και η τεχνική υπηρεσία. Και ενώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 14 υπέρ 15 κατά, αντί για 15 υπέρ 15 κατά, και γι' αυτό παρακαλώ να επαληθευθεί από τη γραμματεία που ήταν η διαφορά στη ψήφο και ή δυνατόν να επαναληφθεί η ψηφοφορία, ίσως και κατά τη διάρκεια ακόμη της σημερινής μας ημέρας, της σημερινής ψηφοφορίας μάλλον, να επαναληφθεί αυτή η ψηφοφορία, στα σημεία στα οποία λόγω του τεχνικού και μόνο προβλήματος, δεν δούλεψε δηλαδή το μηχάνημα, να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Ο πρόεδρος, έχουμε την καταγραφή των ε, ψηφοφοριών από τις τεχνικές υπηρεσίες. Βεβαίως, βεβαίως μπορούμε να επαληθεύσουμε το πρόβλημα αυτό. Θα με ενημερώσετε μέσα σε μερικά λεπτά. Λεπτά, λεπτά. Πριν να κλείσουν οι ψηφοφορίες. Έτσι να έχουμε το περιθώριο να λάβουμε απόφαση αν θα χρειαστεί η επανάληψη της ψηφοφορίας. Είναι σημαντικό το θέμα. Σε μερικά λεπτά παρακαλώ. Can uh, Ωραία, λοιπόν, να σε επανέλθουμε στις ψηφοφορίες. Θα επαναλάβουμε τις ψηφοφορίες εφόσον διαπιστώσουμε ότι υπάρχει λόγος. Ας περάσουμε στο σημείο 22, δεν είναι. Μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ. Ας περάσουμε στο σημείο 22. Εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής. Πρόκειται για μία έκθεση για την εμπορική και επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Μεσογειακό Νότο μετά την Αραβική Άνοιξη με εισηγητή τον Νικολό Ρινάλδη. Ας ψηφίσουμε. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 16 τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές. Εγκρι... Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ 21 Συγγνώμη, υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Κάποιος έχει αντίρρηση. Η προφορική τροπολογία τι είναι. Α, είναι στο παράρτημα. Τη γνωρίζετε λοιπόν. Ας ψηφίσουμε. Τροπολογία 21 με την προφορική τροπολογία ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, επανέλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αυτή ήταν η τροπολογία 21. Ας περάσουμε στην τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 με προφορική τροπολογία. Επίσης βρίσκεται στο παράρτημα. Υποθέτω ότι το γνωρίζετε. Τροπολογία 23 όπως τροποποιείται από την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά 34 υπέρ κατά αποχές εγκρι, απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 40 να συγγνώμη 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 δεν καταπίπτει Α, εγκρίθηκε τροπολογίες τώρα 43 3. Τα έχει ψηφοφορία πρώτο τμήμα ε, υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 λάθος 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 55 με προφορική τροπολογία Α, δεν υπάρχει ε, προφορική τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ συγγνώμη 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 Ελέγχουμε την 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Που ήμασταν στην 65, 64 συγγνώμη, 65 τώρα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 5 και 6 75 και 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία στις αιτιολογικές σκέψεις 1 υπέρ αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τροπολογία 11 κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολόγια 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γνωμοδότηση ΑΦΕΤ ε, η τροπολογία της ΑΦΕΤ ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 καλύπτεται ήδη 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 ε, οι 6 και οι 7 καλύπτονται ήδη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9, 10 ήδη καλύπτονται 11 υπέρ περιμένετε λίγο μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι 6 και οι 7 έχουν εγκριθεί. Ναι. Έτσι λοιπόν καταπίπτει 11, 12 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 13 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πλήρης επιτυχία η τροπολογία της ΑΦΕΤ. Γνωμοδοτή άγκρη, ε, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ανθρωπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ καλύπτεται ήδη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία οκτώ δεν έχει σχέση και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is... Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25 έναντι 5, 0 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Item 23. Σημείο 23. Η Επιτροπή μου ζήτησε να λάβει το λόγο όμως πριν από την ψηφοφορία. Μετά. Όχι πριν. Μετά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τελική ψηφοφορία σε σχέδιο συστάσεως με συγχύτρια με στάκτρια μάλλον την κυρία Κέστιγκερ. Μόνο ναι ή όχι μπορούμε να πούμε, έρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Στάχρη της Χαμοδότησης και την Επιτροπή σας και να επισημάνω ότι το Κοινοβούλιο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ήδη έχει δώσει και την πλευρά του την έγκριση για την συμφωνία. Άρα βαίνουμε ομαλός προς κύρωση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. 24. Μια παράλληλη συμφωνία, πάλι σε διαδικασία έγκρισης, πάλι μια ψηφοφορία, πάλι κυρία Κρίστιγκερ συντάκτης, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε. ομόφωνα και πάλι και συγχαρητήρια στην κυρία Κέστιγκερ. Στο 25 τώρα. Έχουμε τα θέματα τα ήδη διπλής χρήσης με συγκεκριτή τον Πρόεδρο. Σχέδιο σύστασης. Μόνο αυτό έχουμε να εγκρίνουμε υπέρ. Δεύτερη ανάγνωση. Συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 25 υπέρ, μία κατά τέσσερις αποχές. Σημείο 26 άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping εκ μέρου χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Νομοθετικό θέμα. Απλοποιημένη διαδικασία χωρί τροπολογίες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις 27 υπέρ. Καμία ψήφος κατά, τρεις εποχέ. Στο επόμενο βήμα. απλοποιημένη διαδικασία. Άρα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και άρα νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε τις άτυπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Επί τη βάση της μας, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, όπως προβλέπετε, θα έχουμε σε πρώτη ανάγνωση τη συμφωνία. Η πραγματιστική ομάδα, υποφαινόμενος ως πρόεδρος και εισηγητής, με, τις, με διπλή ιδιότητα πλέον, και συντονιστές, στους κυρίους Κάσπαρη, Κάζακ, Στέρντι, Ζαντούα, Σόλτς και Ντάρτμα. Ε, δεν υπάρχουν σκιώδεις εδώ, μόνο συντονιστές. Αν δεν έχετε αντίρρηση, προχωρούμε έτσι. 27. Έκθεση. Έκθεση της πρωτοβουλίας λοιπόν με την κυρία Ντεσαρνή. ανισορροπία, αλλά στο εμπόριο. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών εστερα Τροπολογία 51 καταπίπτει. Πολύ σωστά το επισημάνατε. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται mm. Ας επαληθεύσουμε το 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 54 σε τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών. Τι επαληθεύουμε ακριβώς? Την 57? Να επαληθεύσουμε την 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερευθεί, προφανώς. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Ζαντού. Υπάρχουν αντιρρήσεις προς την προφορική. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε κύριε Ζαντού υπαριθμών 2 προφορική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 59. Με προφορική από τον κύριο Κάσπαρη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. τις ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Και εγκρίνεται. Α επαληθεύσουμε λοιπόν την 59. Ναι, ο καθένας μπορεί να ζητήσει επαληθεύση, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Επαληθεύουμε την 59 και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίθηκε. Ξεκάθαρα. Συμβαστική παριθμών 5 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 64. 64. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπερκατάποχες απορρίπτεται επαληθεύουμε την 154 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε απερίφθη Ποια είναι η επόμενη. Μου βοηθήσετε λίγο. Α, 68. Η 68. Αχα, μάλιστα. Πρώτα είναι 156. 156. Ας ψηφίσουμε την 156 Περ, Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαριστική υπερθμών 6 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 77. Όχι. 75 να ψηφίσουμε μάλλον τώρα, ή, ή, ή το και αυτή. Ψηφίζουμε την 75. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε την 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 20 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Ογδόντα επτά. Ογδόντα επτά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εβδομήντα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπερθμόν 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επόμενο θέμα είναι η 102. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. την 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise number 11 in favor. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποια είναι η επόμενη. 115. Ψήφι 115 τροπολογία. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Εντάξει, να ελέγξουμε την 115. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. οριακά, αλλά απορρίπτεται. 118 τροπολογία. Καλά, δεν τα λέω. 118. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά 120 επαναλαμβάνω την ψηφοφορία ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 120. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οι 121 και 124 τροπολογίες ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 126 υπέρ, κατά. Έχει ζητηθεί έλεγχος. Για ποια. Α, για τις 121 και 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται. Να σκόντε τα χέρια σας. Τροπολογία 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, θέλετε να επαληθεύσουμε. Συμβεβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμ... Όχι συμβεβαστική, απλή τροπολογία. Ποια είναι. Let's move. Και όμως περνάμε σε συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 142. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. 100... Επαληθεύουμε παρακαλώ για την 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. 141. Τροπολογία 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 144 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Οπότε επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πού πηγαίνουμε. Τροπολογία 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφουίζουμε την τροπολογία 19 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με ακούλπα εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Καταπίπτει. Α, πολύ σωστά. Έχετε δίκιο. Επόμενη τροπολογία. 161 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποια είναι η επόμενη. 166. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τι γίνεται με την τροπολογία, μπορείτε να με διαφωτίσετε. Καταπίπτει, παραμένει, Στα σχόλια έχει γίνει ένα λάθος. Καταπίπτει η τροπολογία αυτή. Αντί να λέει ότι καταπίπτει αν εγκριθεί 166, έπρεπε να λέει καταπίπτει αν εγκριθεί 163. Λοιπόν, καταπίπτει. 165 τώρα. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. 167 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτει. Ελέγχουμε. 167 τροπολογία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17. Ψήφι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 174 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 177. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 181. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ κατάποχες, εγκρίνεται. 4 4 Τέσσερα τροπολογία Ψ, ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 τροπολογία υπέρ, Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Όχι, ελέγχουμε το 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία όλα. Συγγνώμη, πάλι έκανα λάθος. Τροπολογία 15, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ Θέλετε να αλλάξουμε την 21 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε την 22 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία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 Μεγάλη πλειοψηφία υπέρ. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Τροπολογία 3. Συμβιβαστική τροπολογία είναι. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46. Δεν πάμε τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Πού πάμε. Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ΔΕΒΕ. ΔΕΒΕ 1. Καβερτκάβερτ καλύπτονται, καλύπτονται που πάμε Δέβε 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέβε 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέβε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέβε 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέβε 18. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 24 υπέρ κατά μισό λεπτό. 23. Για να ελέγξω μισό λεπτάκι αν πρέπει να ψηφίσουμε την 23. Does it fall, does it... Για πείτε μου παρακαλώ αν καταπίπτει ή όχι 23 για να ξέρουμε, να προχωρήσουμε. 156 Καταπίπτει, γιατί έχει κρυθεί 156, άρα περνάμε στην ΤΕΒ 24, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΤΕΒ 26, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΤΕΒ 28, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται Ντεβ 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ντεβ 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Ντεβ 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε, παρακαλώ, την ΤΕΒ 31. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 33 της ΔΕΒ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒ 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νομοδότηση της Επιτροπής Ήτρε που πάμε στην Ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Η 10 έχετε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ήτρε 13. Έχει εγκριθεί. Λίτρο 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή ΙΜΚΟ. Τροπολογία 3 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Για να τσεκάρουμε πρώτα. Μήπως έχει καταπέσει. ψηφίζουμε. Την ύμκο 3. Την ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή Απασχόλησης. Έμπλ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εμπλ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Employment 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία. Ή κάτι μας έχει ξεφύγει. Τελική ψηφοφορία από το σχεδίο γνωμοδότης όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και ο Ντάνιελ Κάσπαρη θέλει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, our, our request would be... εμείς ζητάμε αγαπητοί συνάδελφοι να ψηφίσουμε ξανά για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 30 και για την τροπολογία 40 για την Ευρώπη που είναι αποτελεσματικός προς τους πόρους που έδειξαν αποτέλεσμα 15 προς 40 ενώ συμμετείχαν μόνο 29 μέλη. Για να απαντήσω στο αίτημα του κ. Κάσπαρη για το σημείο 19, δηλαδή τη γνωμοδότηση για την Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία, τρεις ψηφοφορίες, τροπολογίες 14, 30 και 40. Ας ξεκινήσουμε με την τροπολογία 14. Μιλάμε για το σημείο 19 της ημερησία διάταξης. Ε, σχέδιο μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, συζητητής Σαλβατόρε Ιακολίνο. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 14. 14-1-4 της Αλεξανδού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Δεν ήταν κατά τμήματα η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία μόνο για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 30 του Μπερλάνγκε. Μόνο το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία τώρα 40 της Κάθριν Μπιερβέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Χρειάζεται να κάνουμε και τελική ψηφοφορία για το σημείο 19. Σημείο 19 λοιπόν. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε την τελική ψηφοφορία για το σημείο 19. Ο εξοπλισμός ε, του Κοινοβουλίου αρνείται να ε, συνεργαστεί μαζί σας, λέει. Ε, πέρας ψηφοφορία, αστείευεται ο Πρόεδρος, εγκρίνεται με 26 υπέρ, 0 κατά, 4 αποχές, συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή. Item Περνάμε τώρα... So, the vote is... Voting time is closed. Let's... Uh, Πέρας λοιπόν του χρόνου ψηφοφοριών και ας περάσουμε Καταλαβαίνω ότι είστε ανακουφισμένοι που έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε. Σας παρακαλώ, λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, όσοι φεύγετε, παρακαλώ, αναχωρήστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ησυχία. Όσοι παραμείνετε και συζητάτε, παρακαλώ, καθίστε. Okay.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 Okay, let's on. Ε, συνεχίσουμε επόμενο σημείο. Είναι η συμφωνία, εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης απομίμησης. Ο εισηγητής είναι David Μάρτιν της ομάδας των σοσιαλιστών. Έχουμε εγκρίνει ένα χρόνο διάγραμμα το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με τη συνήθη διαδικασία. Δυνατό λόγο στον εισηγητή David Martin. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, η Επιτροπή είχε ένα χρονοδιάγραμμα για το ΑΚΤΑ. Σήμερα θα είχαμε τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Θα είχαμε το σχέδιο έκθεσης για 25-26 Απριλίου και θα ψηφίσουμε σε αυτήν την Επιτροπή στις 30 Μαΐου. Θα θυμάστε ότι ο αρχικός εισηγητής Καντιλαρίφα παρετήθηκε από τη θέση του εισηγητού διότι θεώρησε ότι ήταν υπερβολικά στενό το χρονοδιάγραμμα και δεν προλάβαινε να διεξαγαγεί τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και γενικότερα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τις διάφορες απόψεις που έφταναν στην Επιτροπή όσον αφορά τα δυνατά και τα δύναμα σημεία του ΑΚΤΑ. Στην προηγούμενη συνεδρίαση πρότεινα ένα χρονοδιάγραμμα εναλλακτικό για την αντιμετώπιση της ΑΚΤΑ, που, για το οποίο δεν εξέφρασε κανείς αντίρρηση σε αυτή την Επιτροπή. Ωστόσο, κατανοώ ότι όλες οι ομάδες και ειδικότερα η δική μου ομάδα το έχουν μελετήσει και έχουν μελετήσει το πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα της επικύρωσης ή όχι της ΑΚΤΑ. Οι ομάδες ποιησης ε, που παραπονιόνταν ε, πριν στον προηγούμενο εισηγητή για το χρονοδιάγραμμα, τώρα παραπονιούνται για την παράταση του χρονοδιαγράμματο. Οπότε είναι σαφέ ότι δεν πρόκειται να μείνουν ικανοποιημένοι. Όσοι ήρθαν σε μένα θέλανε η... να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Τώρα θεωρούν ότι αναβάλουμε ε, τη λήψη αποφάσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε λοιπόν με την άκτα. Θυμίζω τους συναδέλφους, ε, στους συναδέλφους γιατί πρότεινα αυτό το χρονοδιάγραμμα και να τονίσω ότι δεν προωθώ το ένα ή το άλλο χρονοδιάγραμμα. Είτε διατηρούμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για ψήφο σε αυτή την Επιτροπή 30 Μαΐου ή υιοθετούμε το άλλο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, ας μην φύγουμε από αυτή την αίθουσα χωρίς να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Η στρατηγική η δική μου βασίζεται σε τρεις πυλώνες να συνεχίσουμε και να κάνουμε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, να ακούσουμε τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών για την άκτα και επίσης να ακούσουμε τις απόψεις των όσων είναι υπέρ της άκτα και να διεξάγουμε δικαινικέ διαβουλεύσεις και συζητήσεις για την άκτα εντός των προθεσμιών που έχουμε στη διάθεσή μας στο δεύτερο κομμάτι στρατηγικής θα ήταν αυτό το κοινοβούλιο να παραπέμψει την άκτα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το σκεπτικό ότι η Κομισιόν ήδη είπε ότι σκοπεύει να το πράξει. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση της Κομισιόν πριν από έξι εβδομάδες ε, όπως φαίνεται θα το είχε, πίστευα ότι θα το έχει παραπέμψει ήδη αλλά όπως φαίνεται θα το κάνει πολύ αργότερα από ό,τι είχα εγώ προβλέψει και έτσι υπάρχει μια απαράδεκτη καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Το σκεπτικό της παραπομπής στο δικαστήριο από το Κοινοβούλιο δεν αποσκοπούσε στην καθυστέρηση της διαδικασίας, αλλά για να κάνουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Εγώ διαφορεύτηκα με τις ομάδες και υπάρχουν συνένεσεις ως προς τις ερωτήσεις που θα θέσουμε στο δικαστήριο σε περίπτωση που ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική. Θα κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις με την Κομισιόν. Το σκεπτικό λοιπόν είναι αυτή η διαδικασία του να λάβουμε μια νομική άποψη δεν καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά από πολύ σαφείς αποφάσεις και ερωτήματα που θέτει το ίδιο το Κοινοβούλιο. Πάντα ήταν σαφέ και το έχω επισημάνει πολλές φορές ε, και σε προηγούμενες επιτροπές, ότι το δικαστήριο το μόνο που μπορεί να μας πει είναι την νομική κατάσταση. Η άκτα χρειάζεται παρόλα αυτά μια πολιτική απόφαση. Σε καμία περίπτωση η γνωμοδότηση του δικαστηρίου δεν αλλάζει την πολιτική απόφαση που θα ληφθεί εδώ. Δεν είναι έτσι σχεδιασμένη η διαδικασία. Θα πρέπει να κρίνει πολιτικά την άκτα το ίδιο το κοινοβούλιο. Ωστόσο, σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θέλουμε να ε, παραπέμψουμε την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα το αφήσουμε να, να το πράξει μόνο η Κομισιόν. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να μην το παραπέμψουμε, Πρέπει να λάβουμε νομική συμβουλή για το κατά πόσο υπάρχει αποτέλεσμα αναστολής ε, λόγω της παραπομπής από την Κομισιόν. Κατά πόσο δηλαδή αναστέλλεται η διαδικασία επικύρωση σε περίπτωση που η Κομισιόν παραπέμψει την άκτα στο δικαστήριο. Δεν είναι σαφές τι γίνεται εάν εμείς σιωπήσουμε θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο αναστέλλεται η διαδικασία η δική μα εντό του ε, Κοινοβουλίου σε περίπτωση παραπομπή από την Κομισιόν. Αυτό το αφήνουμε προ το παρόν στο πλάι. Αυτό πρέπει να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή είναι κατά πόσο εμεί ω Κοινοβούλιο θα πάμε ή όχι στο δικαστήριο. Αρχικά είχε προβλεφθεί αυτή η ε, απόφαση να ληφθεί στην μήνυ Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα. Το δεύτερο μέρο τη στρατηγική όσον αφορά τις δραστηριότητες της ε, Επιτροπής ε, βασίστηκε στο κατά πόσο θα πάμε στο δικαστήριο ή όχι. Δεν ήθελα να υπάρχει νεκρός χρόνος μεταξύ της παραπομπής του ζητήματος στο δικαστήριο και της πολιτικής αξιολόγησης της άκτας στην παρούσα Επιτροπή. Σχέδιό μου λοιπόν ήταν να συντάξω μια ενδιάμεση έκθεση με την οποία θα ζητάω από την Επιτροπή να μας παρουσιάσει λεπτομερώς τη μέτρα υλοποίησης. Είναι σαφές ότι η άκτα αυτή καθεαυτή δεν αλλάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τρόπος όμως υλοποίησης της νομοθεσίας μπορεί να ε, διαστρεβλώσει την φύση αυτής της νομοθεσίας. Αυτό που ρωτάω λοιπόν την Επιτροπή είναι πώς θα υλοποιήσουμε την άκτα, τι υποχρεώσεις θα θέσουμε στους, στις υπηρεσίες παροχής ε, υπηρεσιών διαδικτύου και επίσης θέλουμε να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη αν προβλέπουν ότι Λόγω της ΑΚΤΑ θα τροποποιηθούν τα τοπικά ποινικά δίκαια όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και τις σχετικές παραβιάσεις. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της τελικής πολιτικής αξιολόγησης με που θα ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία. Όπως πολλοί συνάδελφοι και πολλές ομάδες ε, έχουμε την αισθήση σήμερα ότι η καθυστέρηση δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό οτιδήποτε και αν γίνει δεν θα είναι ε, δεσμευτικό από οποιαδήποτε έκθεση από την Επιτροπή. Και οι δημόσιες δηλώσεις της Επιτροπής ε, στο Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θεωρούνται νομικώς δεσμευτικές. Ε, αυτό έχει συμβεί και σε περίπτωση άλλων διεθνών συμβάσεων όπως στην περίπτωση της Καραϊβικής όπου τη συμφωνία είπα Θα εξυπηρετήσει λοιπόν κάποιο χρήσιμο σκοπό η ενδιάμεση έκθεση. Η απόψη μου είναι εάν δεν παραπέμψουμε το θέμα στο δικαστήριο καλύτερα είναι να μην συντάξουμε ενδιάμεση έκθεση και να περάσουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε δύο γύρους, αλλά πριν περάσουμε στο θέμα της ΑΚΤΑ, ίσως οι συναδελφοί θα μπορούσαν να υποδείξουν κατά πόσο ε, υποστηρίζουν την παραπομπή στο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχει τέτοια υποστήριξη, ας ακολουθήσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα και συζητήσουμε ουσιαστικά το περιεχόμενο της άκτα. Ωραία, λοιπόν. Είναι ξεκάθαρο πώς μας τα παρουσιάζει τα πράγματα ο συγητής μένει στην αρχική του πρόταση, ότι δηλαδή θα πρέπει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον το θέμα αυτό πρέπει να το παραπέμψουμε στο δικαστήριο. Αφενός και αφετέρου κατά πόσον θα πρέπει να προβούμε σε μια ενδιάμεση έκθεση με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη καθοριστεί, αντί να συνεχίσουμε τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Οι συντονιστές στη συνεδρίασή τους χθες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμπέρασμα για κανένα από όλα αυτά τα ζητήματα. Συμφώνησαν πάντως να ακούσουν το Συμβούλιο, ότι πρέπει να ακούσουμε το Συμβούλιο. Να ακούσουμε πώς βλέπει το Συμβούλιο τη θέση των κρατών μελών σε σχέση με την ΑΚΤΑ. Διότι είναι μια συμφωνία που δεν χρειάζεται μόνο επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα κράτη-μέλη. Ο εισηγητής βέβαια δικαιούται να επιμείνει να λάβουμε μία απόφαση και για τη δική του έκθεση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν λάβουμε μία απόφαση ως προς αυτό. Διότι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα είναι να συνταχθεί η έκθεση τον Απρίλιο. Άρα δικαιούται να λάβει μια απάντηση ο εισηγητής σε σχέση με αυτές τις δύο προτάσεις, τις οποίες, ε, για τις οποίες μας ζήτησε να λάβουμε μια απόφαση. Είναι δικαίωμα, επαναλαμβάνω, του εισηγητού. Άρα, έχουμε ευθύνε, μην ε, προσπαθούμε να τις αποποιηθούμε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για μένα τουλάχιστον. Ο Ντανίλ Κάσπαρη είναι ο επόμενο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, εμείς στο ΑΛΚΑ, στο ΑΚΤΑ, αισθανόμαστε την ίδια δυσφορία όπω και ο εισηγητή, εμείς στο ΕΛΚΑ. Το ένα θέμα είναι βέβαια το χρονοδιάγραμμα. Σωστά, εχθέ στου συντονιστέ αποφασίσαμε να μην ε, καταλήξουμε σε ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εμείς ως ΕΛΚ προτείναμε πρώτα να ακούσουμε τι έχει να πει το Συμβούλιο στην υπόθεση αυτή. Γιατί σημαντικό είναι για μένα να αφήσουμε αρκετό χρόνο για να κοιτάξουμε την ησυχία μας όλο το θέμα του ΦΑΚΤΑ, όπως πράττουμε εδώ και μερικούς μήνες. Και ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινή γνώμη, γιατί εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, δεν έχουμε αυτό που υπάρχει στις ε, χώρες, σε μια κυβέρνηση με την αντιπολίτευσή της δηλαδή, και ως εκ τούτου δεν είναι ξεκάθαρη οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ομάδων. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν το άκτα καταπολεμά ικανοποιητικά το θέμα των παραποιημένων προϊόντων που ζητούμε και επιδιώκουμε εδώ και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο και ε, με την Επιτροπή τη δική μας αλλά και με τις Επιτροπές Αρμόδιες για Γνωμοδότηση πρέπει να αφήσει αρκετό περιθώριο χρόνου ώστε να εξεταστεί το θέμα εις βάθος. Εμείς τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί ως προς το άκτα τις λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Εμείς το ΕΛΚ. Και θέλουμε να συζητηθεί το θέμα διεξοδικά και με την κοινή γνώμη και με τα κράτη-μέλη και με την Επιτροπή. Επίσης θέλουμε να μάθουμε τι σκοπεύει να κάνει το Κοινοβούλιο, γιατί μου φαίνεται λίγο τυχοδιοκτικό να ξεκινούμε μια διαδικασία όταν δεν είναι τα κράτη-μέλη συνεπή ως προς τα συμπεριφορά τους. Γιατί τα κράτη-μέλη ήταν παρόντα κατά την σύνταξη, κατά την κατάρτιση της σύμβασης άκτα, αλλά ορισμένα από αυτά τώρα δεν προχωρούν σε κύρωση, ενώ έχουν υπογράψει, και αναβάλουν την κύρωση, την κατάθεση της υπογραφής καλύτερα. Επομένω, τώρα δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα ούτε για εμά ούτε για την Επιτροπή. Αν πρόκειται να υπογραφεί ε, αν πρόκειται να γίνει αυτή η υπογραφή ε, στο προσεχές μέλλον. Εκείνοι οι οποίοι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν ξέρουν αν συμφωνούν ή όχι με τη σύμβαση, με τη συνθήκη αυτή. Ε, και εμείς από το Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση, δεν ξέρουμε τι θέση έχουν. Και προφανώς και προσωπικά μπορώ να πω ότι η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται να περιμένει ότι θα να περιμένει να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως και εμεί από πλευρά μα θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πρόκειται να αποφασίσει η γερμανική κυβέρνηση για να την ελέγξουμε. και για να ξέρουν και αυτοί που κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο πράγματι πραγματεύτηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να αφήσουμε χρόνο στην προσοχή μας συνεδρίαση, να καλέσουμε το Συμβούλιο για να ενημερωθούμε πώς βαίνει η κατάσταση και όπως είπα για εμάς το ΕΛΚ που ήδη έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις γιατί δεν μας πείθει το ΑΚΤΑ συνολικά ε, θα περιμένουμε να δούμε εάν καλύφθηκαν οι επιφυλάξεις μας και κυρίως, και κυρίως το θέμα των, ε, της στήριξης της ε, πίστης στο άκτα από πλευράς αυτών ακριβώς που το διαπραγματεύτηκαν. Ένα αυτοί που το διαπραγματεύτηκαν δεν είναι πεπισμένο ότι είναι μια καλή συμφωνία, δεν υπάρχει λόγος να προχωρούμε εμείς σε συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ας δούμε λοιπόν το Συμβούλιο, ας συζητήσουμε μαζί του και, ας συζητήσουμε μαζί του και το θέμα του χρονοδιαγράμματος με την ελπίδα ότι πριν από τις τερινέ διακοπές θα είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε, εφόσον βέβαια δεν προκύψουν νέα στοιχεία από πλευρά του Συμβουλίου, ε, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε στην ανάγκη να επεξεργαστούμε μια ενδιάμεση έκθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπω είπα, αυτοί που το διαπραγματεύτηκαν φαίνεται να μην έχουν πιστεί για το αντικείμενο τη διαπραγμάτευσή του και την αξία του. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμεί στο Κοινοβούλιο πρέπει να χάνουμε χρόνο και να συζητούμε το θέμα αυτό, όταν οι ίδιοι δεν το υποστηρίζουν. Κύριος Μωρέιρα, Πρόεδρε, ε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, κοιτάξτε να σα πω, ο εισηγητή βεβαίω έχει το δικαίωμα να κάνει τι παρατηρήσει ε, και να διατυπώσει τι θέσει του μέσα στην ε, έκθεση του. Δεύτερον, ή συμφωνούμε ότι υπάρχει μια διαδικασία και τη συνεχίζουμε ή αλλάζουμε χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε όμω σήμερα να βγούμε από την αίθουσα χωρί συγκεκριμένη απόφαση. Ή αλλάζουμε χρονοδιάγραμμα ή παίρνουμε σήμερα απόφαση. Πρέπει ο εισηγητή να γνωρίζει τι, με τι είναι αντιμέτωπο. Κύριε Κάσπαρη στα αγγλικά. Πρόεδρε, στα γερμανικά. Στην ημερήσια μας διάταξη δεν αναφέρεται ότι λαμβάνεται απόφαση σήμερα, απλώς ότι συζητούμε τη διαδικασία, ε, δηλαδή μάλλον τη διαδικασία την αποφασίζουν οι συντονιστές. Οι δε συντονιστές εχθές έκαναν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν έλαβαν απόφαση για το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή παραμένει ενισχύ το, το, μέχρι τώρα χρονοδιάγραμμα, για τον Απρίλιο δηλαδή η παρουσίαση της εκθέσεως στην Επιτροπή, του σχεδίου εκθέσεως στην Επιτροπή, με προθεσμία για καθεστροπολογιών στη συνέχεια κτλ. Και δεύτερον, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε σε προσοχή μας συνεδρίαση το Συμβούλιο για να έχουμε το περιθώριο και σε μετέπειτα συνεδρία των συντονιστών να συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αυτό έχουμε συμφωνήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα θέμα να απαντήσουμε σε, στην παρούσα συνεδρίαση στο ερώτημα του εισηγητού, γιατί δεν, μας, δεν το απαιτεί καν το χρονοδιάγραμμα αυτό, ούτε η μερίτσια διάταξη. Πάντω ω προς το χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να δεχθούμε αυτό που προτείνει ο εισηγητή αλλά παρακαλώ και τον εισηγητή να κάνει μια σαφή ε, πρόταση, όπως είχε πράξει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα είχαμε συζητήσει όλα, εμείς είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς πρόταση του εισηγητού. Του ζητήσαμε να κάνει και τις σχετικές προσαρμογές με βάση παρατηρήσεις μας και χθε. Έκλεισε το θέμα της διαδικασίας σε επίπεδο συντονιστών. Δεν υπάρχει λόγο σήμερα να ληφθεί άλλη απόφαση. Η Επιτροπή βέβαια έχει την, ε, απόλυτη, τον απόλυτο έλεγχο του, του χρονοδιαγράμματος, λέει ο Πρόεδρος, και όχι οι συντονιστές. Κύριος Μάρτιν, Πρόεδρε, καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Γκάσπερη, αλλά θα πω το εξή για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ε, έκανα μια πρόταση στην προηγούμενη συνεδρία, δεν την ψηφίσαμε. Η γραμματεία αλλά και εσεί, Πρόεδρε, μου είπατε ότι ω εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα, εφόσον απερίφθη την πρότασή μου, ισχύει το χρονοδιάγραμμα. Εάν δεν αλλάξει λοιπόν το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τώρα σήμερα έχουμε δεύτερη ανάγνωση. Άρα καταθέτω 26-27 Απριλίου το σχέδιο εκθέσεως και θα ψηφίσουμε στι 30 Μαρτίου, Μαΐου. Εγώ πρότεινα να, θα ήθελα μάλλον να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Αλλά αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση σήμερα, χάνεται η ευκαιρία. Με το να μην λάβουμε απόφαση δηλαδή, εγκαταλείπουμε τελείως αυτή την ε, προοπτική, αυτή την, ε, αυτό το ενδεχόμενο. Και συνεχίζω, κάνω εγώ το κείμενό μου, το παρουσιάζω από 25-26 και όπως είχαμε πει αρχικά θα έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πούμε ναι ή όχι στο άκτα, τίποτε περισσότερο ε, και καταλαβαίνω βέβαια ότι οι συνάδελφοι μπορεί να ζητούν περισσότερο χρόνο. Αλλά κοίταξε το άκτα έχει κάνει τόσους κύκλους, το έχουμε δει τόσε φορές. Ήρθε η ώρα πια να διαρρήξουμε αυτόν τον κύκλο και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σλάγκ για, για να αρχίσουμε του υπόλοιπου τονιστέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να καταφερόμεθα κατά του Συμβουλίου ή να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση μεταξύ μας. για τη τελευταία ανάλυση, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε να λάβουμε την πολιτική απόφαση για το αν θα δεχθούμε ή αν θα απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή. Και ως εκ τούτου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξαρτήσουμε την απόφασή μας από την τήρηση ενός προγράμματος. Εάν δεν το Συμβούλιο προτιμήσει να πει ότι θα αποφασίσει μόνο όταν θα έχουμε αποφασίσει εμείς, τόσο το καλύτερο στη τελευταία ανάλυση, γιατί αυτό συνεπάγεται και ενίσχυση της ε, θέσεως του Κοινοβουλίου. Εγώ προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε να επισημάνουμε ξεκάθαρα τις αδυναμίες του συστήματος και βάσει αυτό να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Είπατε και εσείς, Πρόεδρε, ότι υπάρχει ενισχύ χρονοδιάγραμμα ο εισηγητής άλλωστε μας είπε σήμερα και εκείνο ε, τις θέσεις του και μας επέδειξε με τον τρόπο αυτό τη σοβαρότητα με την οποία πραγματεύεται το ζήτημα και πολύ σωστά. Υπάρχουν δηλαδή βάσιμοι λόγοι να χειριζόμαστε με αυτό μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή, αλλά από την άλλη υπάρχει πλέον ένα χρονοδιάγραμμα και πρέπει πλέον να ληφθεί η πολιτική απόφαση αν μας ικανοποιεί το κείμενο ή όχι και αυτό προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στονιστή, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σαφής και ειλικρινής, όχι κοινικός ή εριστικός. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ο εισηγητής έχει το δικαίωμα να ε, λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικέ με την πρότασή του. Επομένω, είτε σήμερα, είτε με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα προβλέψουμε σε προσοχή συνεδρία θα γίνει η ψηφοφορία για την έκθεση. Αλλά δεν ε, μπορούμε να του αρνηθούμε την λήψη αποφάσεως. Έχει δικαίωμα στη λήψη μιας αποφάσεως ο συγκητής. Επομένως, είτε σήμερα, είτε σε, με αλλαγή τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, στην προσοχή συνεδρίαση θα γίνει ψηφοφορία. Γιατί πρέπει να ρηφθεί η απόφαση. Ε, αυτό που δεν μπορώ να δεχθώ και να επιτρέψω είναι να πούμε στον εισηγητή ναι, έκανες μια πρόταση εσύ, αλλά δεν θα λάβουμε σχετικά, σχετική απόφαση σήμερα και για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι σοβαρό αυτό, γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ αγαπητοί συντονιστές, ανταποκριθείτε, απαντήστε συγκεκριμένα στο ερώτημά μου. Είτε ψηφίζουμε σήμερα τα ζητήματα που έχει διατυπώσει ο εισηγητής και στα οποία δικαιούται μια απόφαση, να απαιτήσει μια απόφαση, είτε αποφασίσουμε να αναβάλουμε κατά ένα μήνα το χρονοδιάγραμμά μας, να παρατηρούμε το χρονοδιάγραμμά μας και να πάμε στην προσεχή τακτική ή στους συντονιστές. Ε, χρειάζεται απόφαση από εσά σήμερα και τώρα. Ο κύριος Καζάκ. Πρόεδρε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω το θέμα της νομοδότησης επιτροπής μας. Πρέπει, της ε, έκθεσης επιτροπής μας. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια άποψη, σε μια, απόφαση. Η κατάσταση είναι περίπλοκη ούτως ή άλλως. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η τοποθέτηση των διαφόρων οργάνων. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρχικά υπέρ ε, και πίεζαν και τα κράτη-μέλη για όσο δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση διαπραγμάτευση. Στο μεταξύ όμω εκδηλώθηκε η αντίδραση τη κοινή γνώμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ε, παραπέμψει το θέμα ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πράγμα το οποίο περιπλέκει τα πράγματα ως προς το χρονοδιάγραμμά μας. Όπως ανέφερε και ο κύριος Κάσπαρη. Δεν είναι σαφές το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε επίπεδο Συμβουλίου, διότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία προσυπέγραψαν στο Τόκιο, αλλά απορρίπτουν τώρα την κύρωση της συμφωνίας. Και γι' αυτό νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στον εαυτό μας ως ε, Κοινοβούλιο για να ε, εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη λύση για τη συμφωνία αυτή. Το θέμα είναι αν θέλουμε εμείς να περιμένουμε την απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο κατόπιν, του Δικαστήριο κατόπιν της παραπομπής της Επιτροπής, αν θέλουμε οι ίδιοι ως Κοινοβούλιο να προσφύγουμε παράλληλα στο Δικαστήριο. Εχθές είχαμε την τοποθέτηση νομικής υπηρεσίας. και την υπόδειξη ότι θα ήταν πολιτικά επικίνδυνο το να ε, διατυπώσουμε γνωμοδότηση πριν το δικαστήριο να εκφράσει την ατιμιγορία του. Άρα πιστεύω ότι η δική μας η απόφαση θα ήταν σκόπιμο να αναβληθεί για προσεχή συνεδρίαση, για την προσεχή συνεδρίαση και να ακούσουμε το Συμβούλιο χωρίς βεβαίως να δεσμευόμαστε από αυτό. Ευχαριστώ. Ο Γιάννη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάτι που δεν το πολύ καταλαβαίνω. Απ' τη μία συνεχώς διεκδικούμε ε, την αρμοδιότητα της εξουσίας του Κοινοβουλίου και ε, ξαφνικά, επειδή δεν είναι ξεκάθαρη κατάσταση πουθενά, θα έλεγα, λέμε ότι δεν θέλουμε ούτε να πιέσουμε την Κομισιόν, τα περιμένουμε το Συμβούλιο. Ποια είναι η πολιτική αρμοδιότητα και πολιτική ευθύνη του Κοινοβουλίου. Δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε ένα φάκελο μπροστά μας και έχουμε την ευθύνη να πούμε εάν ναι ή όχι επικυρώνουμε ως κοινοβούλια τη Συμφωνία Άκτα. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση του εισηγητή, ο οποίος πιστεύω ότι έδειξε πνεύμα υπευθυνότητα και κοινού νου. Και μας λέει, υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αυτό το χρονοδιάγραμμα μου λέει ότι εγώ πρέπει να υποβάλλω γνωμοδότηση για το Κοινοβούλιο, όχι η ενδιάμεση έκθεση πλέον, αλλά γνωμοδότηση και νομίζω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την προσέγγιση του εισηγητή και όχι να αρχίσουμε εμείς ως κοινοβούλιο να ε, διαρωτώμεθα κατά πόσο πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι αν υπάρχει ένα κοινοβούλιο κάπου το οποίο θα μπορούσε να κυρώσει μια ευρωπαϊκή απόφαση διότι δεν ψηφίζουμε καμία εμπορική συμφωνία τελικά αν πρέπει επιπλέον να περιμένουμε να επικυρωθεί η συμφωνία στα Εθνικά Κοινοβούλια όλων των χωρών μελών. Τότε σταματάμε και τη δουλειά εδώ πέρα. Εάν έχουμε τη βούληση να έχει ένα κύρο και μια βαρύτητα στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα το Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να περιμένει τρομοκρατημένο και να λέει ότι πω, πω κάποιο μέλο Συμβουλίου θα αλλάξει γνώμη και πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν τελικά εμεί καλά κάνουμε ε, και πηγαίνουμε προ την κατεύθυνση του Συμβουλίου ή όχι. Όχι, εμεί έχουμε πολιτική ευθύνη να γνωμοδοτήσουμε. Ο εισηγητή μα εξέφρασε την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εγκρίνουμε την άποψή του, να την υιοθετήσουμε. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Άρα, τέλη Απριλίου, στην προσοχή μα συνεδρία, θα μα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση του ΟΣΓΙΤΗ μέσω ενδιάμεση έκθεση, μέσω παραπομπή στο δικαστήριο. Θα το δούμε αυτό και ψηφίζουμε το Μάιο την έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, Κύριο Όχι, καλή Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ απόλυτα και αυτό δεν σας κάνει έκπληξη. Εμείς θα θέλαμε μια ενδιάμεση έκθεση. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει ανάγκη για νέο χρονοδιάγραμμα, διότι συμφωνούμε με το γεγονός ε, με όλα αυτά που γίνεται στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο θα πρέπει να το προσαρμόσουμε κάποιος ώστε να συγχρονιστούμε σωστά συμφωνούμε να θέσουμε ερωτήσεις στο Συμβούλιο όσον αφορά το ECJ μπορούμε, μπορούμε να μην αναφερόμαστε καθόλου σε αυτό μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό το θέλουμε υπάρχει, χρειάζεται ένα χρονοδιάγραμμα Ευχαριστώ πρόεδρε Συμφωνώ με εκείνους συναδέλφους που λένε ότι βεβαίως και με πολύ μεγάλη ευσυνητησία πρέπει να ε, παληθεύσει το θέμα αυτό η Επιτροπή μας. Δεν νομίζω ότι κανείς διανοείται να ε, καταχραστεί της ε, περιπλοκότητας της διαδικασίας για λόγους τακτικούς. Εμείς ως βουλευτές εδώ έχουμε καθήκον να υπεραμεινθούμε των δικαιωμάτων, των συμφερόντων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή να έχουμε αφοσιωθεί και πρέπει να εξετάσουμε τον φάκελο αυτών του άκρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τηρηθεί επακριβώς το χρονοδιάγραμμα και για να απαντήσω στην ερώτησή σας έχουμε συζητήσει εξωτικά το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας, στην ομάδα μας και πιστεύουμε ότι ως Κοινοβούλιο δεν πρέπει να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά να επιτελέσουμε το έργο μας και να τοποθετηθούμε προ το πολιτικό ζήτημα που είναι αυτό της εξέτασης της συμφωνίας. και της καταγραφής των θετικών και αρνητικών σημείων της ε, συμφωνίας, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο διατάφτα. Βεβαίως, το να γύρει μια συζήτηση, μια ακρόαση μάλλον με το Συμβούλιο, δεν είναι απαραίτητα τόσο περιττό. θα ήταν καλό να δούμε γιατί τα κράτη-μέλη, ενώ είχαν καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και είχαν καταλήξει μια συμφωνία, τώρα ξαφνικά δεν τολμούν να την κυρώσουν. Τι είναι αυτό που τα τρομάζει τόσο. Είναι κάτι το οποίο εμεί ω Κοινοβούλιο θα ήταν σκόπιμο να δούμε. Ίσως και άλλε συμφωνίε ή ρυθμίσει στον ευρωπαϊκό χώρο, οι οποίε έχουν να κάνουν με κάποιες πτυχές του άκτα και είναι εκκρεμή στο πεδίο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστούν με το πεδίο αυτό, με το πνεύμα αυτό γιατί θα έχουμε και προσεχή γύρω ε, για τελωνιακές διατάξεις, για ε, αγαθά που έχουν να κάνουν με την πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Ε, θα έχουμε να κάνουμε με διάφορες σχετικές διατάξεις και γι' αυτό καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε καλά αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συναδέλφοι. Καθήκον μου είναι να φροντίζω για την τήρηση των κανόνων. Τα δικαιώματα του πρέπει να τηρούνται. Οι προτάσεις του ισχύουν. Έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για αυτές. Δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση με σχέδιο έκθεσης διότι όπως ανέφερε πριν ληφθεί απόφαση παραπομπή στο δικαστήριο ή σε περίπτωση που ληφθεί ε, απόφαση για παραπομπή στο δικαστήριο τότε θα χρειαστούμε ενδιάμεση έκθεση. Όπως βλέπω η σε περιπτωση που ληφθει αποφαση για παραπομπη στο δικαστηριο τοτε θα χρειαστουμε ενδιαμεση εκθεση οπως βλεπω η η επιτροπη δεν, οι ομάδες και η επιτροπή δεν είναι έτοιμοι να ψηφίσουν σήμερα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αναβάλουμε την απόφασή μας. Η επίσημη μου πρόταση είναι να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα, κατα, το μετατοπίσουμε κατά ένα μήνα, ώστε να αποδεσμεύσουμε τον εισηγητή από την υποχρέωσή του να παρίσταται στην επόμενη συνεδρίαση και να παρουσιάσει μια, ένα σχέδιο έκθεσης ε, για τη συνένεση. Αυτή είναι η επίσημή μου πρόταση προς εσάς. Η Επιτροπή ελέγχει το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει, κατά την ανάποψή μου, να λάβει μια απόφαση. Κάσπαρη. Ε, Επανέρχομαι, Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση. Στην τελευταία συνέδρια της Επιτροπής μας, ο εισηγητής είχε προτείνει να κάνει την ε, πρόταση για κοινή από τη Επιτροπής μας πάρα πολύ του θέματο στο δικαστήριο. Το συστήσαμε πολύ μεταξύ μα και στην Επιτροπή. Κατέστη το μεταξύ σαφέ, κατέστησαν μάλλον σαφεί οι προτάσει τη Επιτροπή. και μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κανεί με συγκεκριμένη πρόταση για παραπομπή στο δικαστήριο. Γι' αυτό το λόγο δεν βλέπω γιατί πρέπει να τοποθετηθούν οι ομάδε, αφού κανεί δεν ζητεί την παραπομπή στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει λόγο. μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Και για το χρονοδιάγραμμα ε, ορίζει ήδη ότι θα καταθέσει ο εισηγητής το σχέδιο εκθέσεως τον Απρίλιο, θα οριστεί προθεσμία για ψηφοφορίες, θα γίνει ψηφοφορία, μετά θα πάει στην Ολομέλεια και επίσης επιτρέψτε μου σε αυτό βαθμό να αποκαλύψω τα όσα συζητήθηκαν χθε στους συντονιστές. Δεν άλλαξε τίποτα ως προς το χρονοδιάγραμμα γιατί δεν ελήφθη καμιά απόφαση από τους συντονιστές. Εφόσον ελήφθη καμιά απόφαση ισχύουν τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Δηλαδή προσκαλούμε το Συμβούλιο σε προσεχή συνεδρίαση και σε μεταγενέστερη συνεδρίαση των συντονιστών εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από το Συμβούλιο, μπορεί να ξανασυζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν είναι θέμα το οποίο χρειάζεται συζήτηση. Δεν χρήσιστε ίσως η διαδικασία του χρονοδιάγραμμα, εφόσον ήδη είναι σαφή. Έχουμε στην, ε, στο πρόγραμμά μας την κατάθεση του σχεδίου εκθέσεως τον Απρίλιο, μετά έχουμε τις τροπολογίες ε, και την ψηφοφορία το Μάιο και μετά πάμε στην ε, όλο μέλη, εφόσον θα έχουμε ήδη μεταξύ το περιθώριο να συζητήσουμε και το, με το Συμβούλιο και να δούμε και τα αποτελέσματα της παραπομπής, τη απόφαση περί παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι η εικόνα θα είναι πλέον σαφής. Και νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Αν δεν λάβουμε κάποια διαφορετική απόφαση σήμερα, σημαίνει ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, λαμβάνουμε την απόφαση να μην, να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό συναπάγεται η μη λήψη αποφάσεω. Δεν βλέπω κανένα αίτημα μέχρι στιγμή ε, για ενδιάμεση έκθεση από πλευρά του εισηγητού, άρα ούτε αυτό χρειάζεται να συζητηθεί. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλη αυτή η αναστάτωση έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους οι, οι ομάδες. Εγώ τουλάχιστον από πλευρά της ομάδας μου επισημαίνω ότι πολλά από τα ερωματικά που μας απασχολούν δεν έχουν ακόμη απαντηθεί και ως εκ τούτου θα ήταν καλό να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις γιατί έτσι θα διευκολυνθεί και η ε, επιλογή μιας απόφασης από πλευράς μας. Όπως καταλαβαίνω η Επιτροπή αυτή μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε ημερολόγιο οποτεδήποτε. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Εάν εγώ αποφασίσω να για την ψηφοφορία, να αλλάξω το ημερολόγιο, να αλλάξω την ημερομηνία ψηφοφορία, η πλειοψηφία τη Επιτροπή αυτή μπορεί να το αποφασίσει. Όπω κατάλαβα εγώ, ο εισηγητή παρουσίασε τις ιδέες του στην προηγούμενη συνεδρίαση και δεν έχει αλλάξει γνώμη ότι πρέπει να ψηφίσουμε για δύο πράγματα κατά πόσο θα το παραπέψουμε το ζήτημα στο δικαστήριο δεύτερον κατά πόσο θα συντάξουμε μια ενδιάμεση έκθεση έχει το δικαίωμα να ζητήσει τέτοια ψηφοφορία δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε παραβιάζουμε τα δικαιώματά του εάν τον αναγκάσουμε να δημιουργήσει σχέδιο σύστασης για συνένεση ενώ αυτό προτιμά μια ενδιάμεση έκθεση. Έχει λοιπόν το δικαίωμα είτε αποσύρει την πρότασή του, είτε για λόγους ε, δικαιοσύνης θα πρέπει να ψηφίσουμε κατά πόσο θα αναστείλουμε το ημερολόγιο κύριε Σίγητα. Ήθελα να πω ας είμαστε σαφείς αλλά τίποτα δεν είναι σαφές όσον αφορά το, την άκτα. Όσον αφορά την παραπομπή στο δικαστήριο, πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε απόφαση τώρα και να την αναφέρουμε στην Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα. Γιατί αν την αναστείλουμε, αν αποφασίσουμε να συντάξουμε κάποιο ψήφισμα για την Ολομέλεια του Μαΐου ή του Ιουνίου, μετά οι νομικές υπηρεσίες πρέπει να εξετάσουν την πρόταση και μετά θα έχουμε και άλλη καθυστέρηση και μιλάμε για μια δικαστική υπόθεση που θα διαρκέσει 18 μήνες. Αυτή εδώ η 7η ε, θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει την άκτα. Δεν πρέπει να περάσει αυτό το θέμα στο επόμενο, στο επόμενο κοινοβούλιο το 2014. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να λάβουμε απόφαση τώρα και να πάει στην Ολομέλεια την Πέμπτη. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε η πρότασή μου για παραπομπή στο δικαστήριο αποσύρεται και έτσι δεν βλέπω για ποιο λόγο σε τέτοια περίπτωση να συντάξω και ενδιάμεση έκθεση. Μπορώ να περάσω στο αρχικό χρονοδιάγραμμα και να ε, δημιουργήσω μια σύσταση στην οποία θα ψηφίσετε με ναι ή όχι. Τα πράγματα λοιπόν είναι σαφή. Ζητώ από αυτή την Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσο σύμφωνα με αυτή την πρόταση του εισηγητού θα ψηφίσουμε τώρα για το αν θα έχουμε παραπομπή στο δικαστήριο ή όχι. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Παρακαλώ μην εκνευρίζεστε κύριε Κασπαρή. Είμαι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία σε αυτή την Επιτροπή. Μην προσπαθείτε να προεδρεύσετε στη θέση μου. Θα ρωτήσω αυτή την Επιτροπή κατά πόσο πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι για το ζήτημα της παραπομπής αυτού του ζητήματος στο δικαστήριο. Εάν απαντήσουμε όχι, ε, εάν πούμε ναι, η δεύτερη ψηφοφορία θα, είναι, θα αφορά το κατά πόσο αυτή η Επιτροπή θέλει ολομέλεια να παραπέμψει αυτό το δικαστήριο στο δικαστήριο. Έχουμε λοιπόν δύο ψηφοφορίες. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε σήμερα για το κατά πόσο θα παραπέμψει αυτό το ζήτημα στο δικαστήριο ή όχι, κύριε Κάσπαρη. Ε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής έκανε μία πρόταση ο εισηγητής ε, για παραπομπή στο δικαστήριο. Πολύ καλά. Και προφανώς αυτό επαναλαμβάνει τώρα και ο εισηγητής. Αλλά δεν υπάρχει γραπτό αίτημα για παραπομπή στο δικαστήριο και πάντοτε στην Επιτροπή μας ε, συνηθίζουμε να ψηφίζουμε ε, πάνω σε γραπτές προτάσεις και όχι σε προφορικές μέσα σε συνθήκες πίεσης. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεύτερον, το ζήτημα περί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν προβλέπεται στην ημερησία μας διάταξη. Την ορίσαμε δε εμείς εχθές ε, ξεκάθαρα στην αρχή της συνεδρίασης και σας διαβεβαιώ ότι εγώ δεν έχω εκνευριστεί καθόλου. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος γιατί γνωρίζω όλες τις τοποθετήσεις και εκείνων βεβαίω που έχουν πει ότι ίσως να ήταν καλό να πάμε στο δικαστήριο αλλά δεν έχει κατατεθεί πρόταση για να πάμε στο δικαστήριο και εφόσον δεν προβλέπεται και μέσα στην ημερησία μας διάταξη δεν υπάρχει θέμα για ψηφοφορία στην ε, ε, διάρκεια της παρουσίας συνεδρίασης. Δεν καταλαβαίνω, ίσως κάτι, ίσως κάτι να έχω μπερδέψει, αλλά δεν βλέπω καμία γραπτή πρόταση για την παραπομπή στο δικαστήριο. Ακόμα και αν το προτείνει ο Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο εκνευρισμού, ούτε είμαι εκνευρισμένος εγώ ο ίδιος. Άλλωστε θα πρέπει να επισημάνω ότι τα προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει εμεί έχουμε βρει εμεί στο θέμα του άκτα όπω και οι άλλε ομάδε, είναι προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να λύσει το δικαστήριο. Δεν θα μα λύσει κανένα πρόβλημα δηλαδή η παραπομπή. Όσον αφορά τον τρόπο του αιτήματο, ε, αυτά είναι αρκετά Ακριβεί προτάσει. Δεν υπάρχει λόγο για έγγραφη πρόταση κατά την άποψή μου. Περνάμε λοιπόν. Ο κύριο David Μάρτιν. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να περιπλέξω κι άλλο τα πράγματα. Να προτείνω μια διαδικασία δύο σταδίων. Ψηφίζουμε τώρα για το κατά πόσο θέλουμε να γίνει ψηφοφορία και αν υπάρχει βούληση για ψηφοφορία μπορούμε να ψηφίσουμε στις 3. Έχουμε ήδη μια, ένα σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για την παραπομπή στο δικαστήριο. Το έχουν την έχουν δει όλες οι ομάδες και έχουμε δηλαδή αυτό το κείμενο για το οποίο μπορούμε να ψηφίσουμε στις τρεις. Αλλά ας ψηφίσουμε πρώτα για το κατά πόσο θέλουμε να ψηφίσουμε. Και αλλιώς, εάν η απάντηση είναι όχι, κλείνει το ζήτημα. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για το κατά πόσο θα ψηφίσουμε για την παραπομπή σήμερα το απόγευμα. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι. We'll have a vote Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Η ερώτηση είναι ποιος είναι υπέρ του να ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα επί της προτάσεως του εισηγητή για παραπομπή αυτού του ζητήματος στο δικαστήριο. Δεν ψηφίζουμε επί του περιεχομένου, ψηφίζουμε για το κατά πόσο πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό σήμερα το απόγευμα. Είναι σαφές? Аз, извинявайте, господин председател, явно нещата станаха доста сложни. А, доколкото разбрах доклад... Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται να έχει περιπλακεί η κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτά που λέει ο εισηγητής θα ήθελε να ληφθεί απόφαση σήμερα για το κατά πόσον μπορούμε να ε, λάβουμε απόφαση για πιθανή, να ψηφίσουμε δηλαδή για πιθανή παραπομπή στο δικαστήριο. Και αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, μας λέγει ο εισηγητής ότι δεν θα σημαίνει ότι δεν θα παραπέμψουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την υπόθεση. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η απόφαση αυτή μπορεί να αναβληθεί για την προσεχή συνεδρίαση. Όμως ο εισηγητής μας λέει ότι αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, εγκαταλείπει την πρότασή του για παραπομπή στο δικαστήριο. Εάν δεν ψηφίσουμε σήμερα, αυτό θα συνεπάγεται και αναβολή για την προσεχή συνεδρίαση της προφορίας ή όχι. Κύριο Ζαντό. Δεν καταλαβαίνω πώς εμείς μπορούμε να κάνουμε παραπομπή στο δικαστήριο όταν δεν γνωρίζουμε σήμερα σε ποια βάση και σε ποιο βαθμό θα ε, πραγματοποιήσει παραπομπή η Κομισιόν. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Ε, προσπαθούμε να πάρουμε αποφάσει για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που έχουμε στα χέρια μα είναι ένα ημερολόγιο και την ευθύνη του εισηγητή την ευθύνη να μας δώσει μία, όχι ενδιάμεση έκδοση, αλλά ένα σχέδιο ε, γνωμοδότησης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί να κάνουμε ψηφοφορία σήμερα σε σχέση με όλα αυτά. Περνάμε σε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έχει ως εξή. Παρακαλώ. Ποιος φοβάται την ψηφοφορία. Αφήστε να αποφασίσει η Επιτροπή. η ουσία, το θέμα είναι το εξή. Ποιο είναι υπέρ του να διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα, όπως το ζήτησε ο εισηγητή για το κατά πόσο πρέπει να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να παραπέμψει το ζήτημα στο δικαστήριο. Φύζουμε τώρα. Yes, yes, Yes. Uh, so my question is just... Ε- η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν αυτή τη στιγμή, όπως επιθυμεί ο εισηγητής, ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε σήμερα επί του ζητήματος στις 3 η ώρα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο εισηγητή, ότι ταυτόχρονα ψηφίζουμε ουσιαστικά κατά της παραπομπής του θέματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σωστά. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, όλοι μπορούν να κάνουν την ίδια πρόταση ανα πάσα στιγμή. Παρακαλώ μην μπερδεύετε τα πράγματα ο εισηγητής έχει το δικαίωμα να θέσει τους όρους στη δική του πρόταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν ψηφίσουμε τώρα ότι δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία το απόγευμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποια πρόταση στο μέλλον. Συνεπώς σας παρακαλώ μην μπερδεύετε τα πράγματα. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν έχω καταλάβει. Τελώ υποσύγχυση αυτή τη στιγμή και θέλω την συμβουλή σας. Εγώ είμαι κατά της προσφυγής στο δικαστήριο, αλλά κατά και της ενδιάμεσης έκθεσης. Είμαι υπέρ της λήψης άμεσης απόφασης. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Please, Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν είναι αστεία πράγματα. Ε, το θέμα είναι σοβαρό. Λοιπόν, μιλάμε για ψηφοφορία σε δύο φάσεις. Δύο ε, σκέλη, αν θέλετε. Το κατά πόσον θα παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ή όχι, αυτό θα το αποφασίσουμε το απόγευμα, ανεξαρτήτως της θέσης σας ε, του κατά πόσο θέλετε να προσφύγουμε ή όχι στο δικαστήριο, αυτό δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την πρώτη ψηφοφορία που θα έχουμε. Δηλαδή, να αποφασίσουμε το απόγευμα ή με άλλο τρόπο ή άλλοτε. Any other request. Λοιπόν, δεν πρόκειται να δεχθώ άλλα αιτήματα. Δεν θέλω να δώσω το λόγο σε κανέναν άλλον. Σας είπα πριν ότι θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας παρακαλώ λοιπόν να ψηφίσετε ως προς το εξής. Ποιος είναι υπέρ να ψηφίσουμε το αίτημα του εισηγητού σήμερα το μεσημέρι. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ, για σηκώστε τα χέρια. Ποιοι είναι υπέρ. Ωραία, ας κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Βάλτε τις κάρτες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, ναι, Γαντάνιελ Κάσπαρη, παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, λέει ο κ. Κασπαρή, αν η πλειοψηφία υπερψηφίσει το να γίνει ψηφοφορία το μεσημέρι, πείτε μας σας παρακαλώ, τι θα ψηφίσουμε, ποιο έγγραφο θα ψηφίσουμε. Μα όλα αυτά αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε διαδικασία υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο να ψηφίζουν, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τηρείται ο κανόνα για τι γλώσσες, είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοια πρεμούρα, γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Δεν δέχομαι μετά από τρία χρόνια στην Επιτροπή αυτή δεν δέχομαι να αρχίσουμε να αλλάζουμε την μέση διάταξη στις συνεδριάσεις. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ε, σε καμία περίπτωση διατεθμένος να δεχθώ κολλησιεργίες. Όταν έχουμε ε, την ανάγκη να ψηφίσουμε για κάποιο θέμα. Λοιπόν, το μεσημέρι είναι ξεκάθαρο ότι θα ψηφίσουμε. Το είπε και ο συγητής, το ξεκαθάρισε. Λοιπόν, α σοβαρευτούμε λιγάκι παρακαλώ και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Μέρφυ. Όχι, έχω ζητήσει το λόγο. Όχι, λέει ο πρόεδρος, δεν πρόκειται να ξαναδώσει το λόγο σε κανέναν. Ο κύριος Μέρφυ. όχι, και εμείς έχουμε δικαίωμα να λάβουμε το λόγο. Πρόεδρος, όχι, δεν πρόκειται να δώσει το λόγο σε κανέναν αν δεν ψηφίσουμε πρώτα. Δεν δίνω σε κανέναν το λόγο, δεν δέχομαι να κολλησιεργεί κανένας εδώ στην Επιτροπή πλέον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Έκλεισα την ψηφοφορία. Εγκρίνεται αυτό. Δηλαδή, θα ψηφίσουμε το μεσημέρι την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Let's move to item 29. Και τώρα περνάμε στο σημείο 29.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 There Κυρίες και κύριοι. Mr. President. There is an item left. Έχει μείνει ένα σημείο για την για διάταξη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν περισσότερα πράγματα. Δεν υπάρχει μόνο η άκτα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το σημείο 29, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε. Ο Ιούλιου Βίνκλερ είναι ο εισηγητής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δικαιούται να τον ακούσουμε ο εισηγητής. Έχετε το λόγο κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι βέβαιος ε, αν ε, κανείς ενδιαφέρεται να ακούσει αυτά που έχω να πω και πόσο χρόνο έχουμε. Αλλά τέλος πάντων σας ευχαριστώ για αυτή τη ε, δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω στην συντομία κάποιες από τις ιδέες μου για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στις χώρες μας ε, αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέμα με την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, να, γίνουν να, ε, να παγκοσμιοποιηθούν λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ούτως ή άλλως αντιστοιχούσαν 99% των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενιαία αγορά, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι τόσο φιλική ε, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, μία στις τέσσερις ΜΜΕ έχει δραστηριότητα εκτός των εθνικών συνόρων κατά την τελευταία τριετία βάσει των στοιχείων που έχουμε λάβει ε, από στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ε, εμπορεύονται ή επενδύουν μόνο ε, στην εσωτερική ένωση αλλά και εκτός ε, των φυσικών συνόρων της Ένωσης. Εάν δούμε, ή μάλλον πώς να το πω, αν αναλύσουμε το διεθνές εμπόριο με τρίτες χώρες, είναι ακόμα πιο αδύναμες οι επιδόσεις. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, διαπίστωση στο το 13% μόνο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ένωση δραστηριοποιούνται και σε αγορές εκτός Ένωσης. Πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν. Πρώτα απ' όλα για να βελτιώσουμε τις εμπορικές, ε, τους εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορούν σε κάποιο βαθμό όλε να δραστηριοποιούνται διεθνώς. Δεύτερον, πρέπει να καταπολεμηθούν οι γνωστοί φραγμοί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια που αποτρέπουν τις μικρομεσαίε επιχειρήσει ακόμη και από το να σκεφτούν ε, να προβούν σε διεθνή δραστηριότητα. Και ένα άλλο, κομμά, ένα άλλο στοιχείο το οποίο περιλαμβάνεται και στην ανακοίνωση τη Κομισιόν είναι η χαρτογράφηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό των σχεδίων στήριξης, ε, εθνικής στήριξης που παρέχεται από τις δημόσιους ε, ε, φορείς και από την επιχειρηματική κοινότητα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν θα μπορούσαν να προβαίνουν σε εξαγωγές. Αυτό όμως δεν είναι επαρκές. Στην Ευρώπη υπάρχουν ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να τις αναλύσουμε, δηλαδή μέγεθος, δραστηριότητα, προέλευση και ιστορικό των επιχειρήσεων. Θα θέλαμε να ξέρουμε και τι θα συμβεί μετά τη χαρτογράφηση που μας λέει η Κομισιόν ότι θα πράξει. Θα χαρτογραφήσει δηλαδή αυτά τα σχέδια, τα προγράμματα στήριξης, αλλά ποιο είναι το επόμενο βήμα. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν θα συνεχίσω μέχρι ότου σταματήσουν τα πηγαδάκια. Okay, uh, thank you, uh, uh, information... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να κλείνουμε, θα πρέπει να δίνονται με πιο προσβάσιμο τρόπο οι πληροφορίες, ενώ υπάρχει και ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ε, φορέων στι τρίτε αγορέ και θα πρέπει να ορίσουμε ποιε είναι οι αγορέ προτεραιότητα. Η Κομισιόν στην ανακοίνωσή τη έχει ένα κατάλογο χωρών. Αν δούμε αυτόν τον κατάλογο, Μπορούμε να φανταστούμε ότι αν ε, κάθε επιτροπή, ε, η επιτροπή προτείνει την Ουκρανία, α πούμε, γιατί δεν προτείνει και τη Μολδαβία. Εάν έχουμε τι ευρωμεσογειακέ χώρες, γιατί να μην έχουμε και από τα Δυτικά Βαλκάνια κάποιες χώρες σε αυτόν τον κατάλογο. Πολύ σύντομα ήταν αυτές κάποιες ε, σκέψεις για τον κατάλογο των χωρών που περιλαμβάνει η ανακοίνωση της Κομισιόν. Η μόχλευση τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ω στόχο, είπαμε, την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι τη ανακοίνωση είναι κάπω απογοητευτικό για να είμαι και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ανησυχούν τι μικρές επιχειρήσει, αλλά τα οποία δεν λαμβάνονται και τόσο υπόψη στην εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό συζητείται εδώ και καιρό. Υπάρχει ένας κατάλογος δράσεων, είπαμε η κατάργηση των εμπορικών φραγμών, φιλική νομοθεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, βελτιωμένη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες προμήθειε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά τα προτείνει και η Κομισιόν, αλλά δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο, τι εργαλεία ε, θα υπάρξουν για την πρόθεση όλων αυτών των στόχων. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και εν κατακλείδη, επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντική ανακοίνωση αυτή, έχει μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Εμεί ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα πρέπει να αναστρέψουμε την ε, πυραμίδα αυτή. Θα πρέπει η προσέγγιση να είναι πιο πολύ από κάτω προς τα πάνω. Θα κάνουμε λοιπόν τις τροπολογίες μας, θα έχουμε και βέβαια τη συζήτηση με τους συναδέλφους για να βελτιωθεί η έκθεση. Θα ακούσω με μεγάλη προσοχή όλα τα σχόλια των συναδέλφων. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Και τώρα περιμένω να ακούσω με ανυπομονησία τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Όπως προείπα αυτή η γνωμοδότηση είναι για την Ήτρε. που βασιστεί στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν για τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Ε, Τζαν Λούκα, σου έχεις το λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Έχουμε εμείς συνηθίσει εδώ και καμποσό καιρό από τότε που υιοθετήθηκε το Small Business Act έχουμε συνηθίσει να θέτουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας ε, και διάφορα επιχειρήματα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ακόμη και την εποχή με την ύφεση, ειδικότερα σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, ε, υποστηρίζουμε την οικονομία βάσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παίζουν μεγάλο ρόλο και για την απασχόληση πέραν των ωφελών που δεν έχουμε καταφέρει να αποκομίσουμε σε αυτό το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι η μικρομεσαία επιχείρηση βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάσταση των επιμέρου ατόμων, ειδικά όσων υποφέρουν περισσότερο αυτή τη δύσκολη εποχή. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αντί να κοιτάμε τις πολιτικές, Εμεί κοιτάμε ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις του τι είναι απαραίτητο να κάνουμε, ε, αλλά ο κατάλογος των πραγμάτων πρέπει να κάνουμε δεν υποστηρίζεται πάντα από πολιτικές επιλογές ή από νομοθετικές επιλογές. Ακόμη και ο προσανατολισμός των κονδυλίων δεν γίνεται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τίθενται ερωτήματα που αφορούν τους κανόνες διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των κοινοπραξιών εξαγωγών, κοινοπραξιών για την προμήθεια πρώτων αλλά και ε, των συστημάτων που θα μας προστατέψουν από επιθέσεις όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, ειδικότερα στις χώρες όπου είναι πιο δύσκολη η διείσδυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προστασία η διαφύλαξη της ποιότητας των προϊόντων τους. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανωθεί ώστε να εξοπλιστεί με καλύτερους κανόνες που όχι μόνο θα αποσκοπούν στο να υπάρχουν περισσότεροι κανόνες αλλά και στην απλούστευση. Λίγοι κανόνες σαφείς που εξαλείφουν ε, τα, τα μη δεσμολογικά εμπόδια που εμποδίζουν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν σε άλλες χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπαμε και προηγουμένως μιλώντας για τη σχέση με την Κίνα. Επίσης χρειάζεται να υποστηρίξουμε τη δραστηριότητα των ΜΜΕ με επαρκή κίνητρα, όχι με υπαρξιακές πολιτικές, με πολιτικές κινήτρων που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη στους στρατηγικούς τομείς. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και προς τις, ανταγωνιστικές, προς τις αναδυόμενες οικονομίες. Μην ξεχνάμε ότι μπορούμε ακόμη να συνεχίσουμε να είμαστε βιομηχανία του κόσμου. Εδώ και κάποια χρόνια είμαστε το γραφείο του κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους τομείς τους οποίους θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας που σχετίζονται με ένα άλλο σύστημα ποιότητας. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είτε η αναθεώρηση του SBA είτε η ανακοίνωση της Κομισιόν πρέπει να, και η ανακοίνωση της Κομισιόν πρέπει να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πολιτικές που θα προκύψουν πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες από αυτές που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Διατηρούμε λοιπόν μια επιφύλαξη μέσω των τροπολογιών θα θέλαμε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε περισσότερο τους στόχους που έχουμε θέσει ώστε να αποφύγουμε να έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο πραγματών που θέλουμε να κάνουμε χωρίς ε, να ε, δημιουργήσουμε νέα μέσα πολιτικά, νομικά και οικονομικά ώστε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο. Ας ακούσουμε την Κομισιόν. Διότι σε τελική ανάλυση όλο αυτό αφορά μια ανακοίνωση της Επιτροπής. Please is Could you yes. tell Θα μας πείτε και το ονοματάκι σας. Χρήστος Κυριάτης από την DG Enterprise της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και ιδιαίτερος σημειώνουμε και εκτιμούμε τα σχόλια του συγητού και των λοιπόν μελών της Επιτροπής, όπως γνωρίζετε ήδη. Μας απασχολεί αυτή η επιχείρηση καταγραφής, χαρτογράφησης των επιχειρήσεων, ώστε να δούμε και πώς οι φυστάμενες υπηρεσίες στήριξης σε επίπεδο μελών μπορούν να καταστούν και πιο ορατές ώστε να προσεγγίσουν τον πελάτη που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση και επίσης ώστε να αναζητηθούν και καλύτερες συνεργασίες μεταξύ των υφισταμένων είδη υπηρεσιών ή να εντοπιστούν κενά, στα οποία θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλάβουμε δράσεις συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις των εθνικών αρχών, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών. Πιστεύουμε, μάλλον εργαζόμαστε έτσι ώστε να μην περιοριστούμε μόνο σε ένα ευχολόγιο, αλλά να προσδιορίσουμε πολιτικές Αποτελεσματικέ. Ξέρετε ήδη ότι υπάρχουν πολιτικέ που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η παραδείγματι η προσπάθεια για την κατάργηση των φραγμών στο εμπόριο μέσα από την Συμφωνία TVT του ΠΟΕ η δουλειά που γίνεται προς την πρόσβαση στις αγορές από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δουλειά που γίνεται στην τυποποίηση και που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή η δουλειά που έχει να κάνει με τον έλεγχο ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των πολιτικών μας. Επίσης έχουμε μια σειρά διατάξεων μέσα στο τωρινό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και επίσης μέτρα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν αυτές επιδιώκουν να βγουν στη διεθνή σκηνή. Το πρόγραμμα COSME, ανταγωνιστικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσεται στο προσεχές δημοσιονομικό, πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020 και μέσω όλων αυτών των δράσεων πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα ε, επιχειρηματικό πλαίσιο πρόσφορο για ανάπτυξη επιχειρηματική δραστηριότητα και εύχριστο για τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε τη θετική ανταπόκριση από πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ο δε ρόλο μας είναι να προσδώσουμε περισσότερη ορατότητα σε αυτές τις υπηρεσίες και όχι να επαναλάβουμε τα όσα ήδη πράττουν τα, σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, αν ε, υπάρχει ανάγκη, στηρίζουμε και μικρομεσαιες επιχειρήσεις από άλλα κρατημέλη, γιατί όντως υπάρχουν κρατημέλη τα οποία δεν προσφέρουν αρκετή υποστήριξη στις επιχειρήσεις τους, αυτές θέλουν να βγουν στο διεθνές πεδίο. Επίσης, χώρες προτεραιότητας. Υπάρχει ένας ενδεικτικός κατάλογος. Γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταρχάς αναπτύσσουν δραστηριότητες ε, σε εθνικό επίπεδο, άρα είναι τοπική η δραστηριότητά τους, μετά ανοίγονται σιγά σιγά προς τη γειτονία τους και όπως είπε και ο συγητής, βεβαίως η Ρωσία, η Ουκρανία αναφέρονται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να στραφούμε και προς άλλες χώρες όπως η Μολδαβία που αναφέρατε ή άλλες χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βίγκλερ, θέλετε να πείτε δύο λόγια για να κλείσει το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους συναδέλφους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρεις σύντομες ιδέες. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω πως αντιλαμβάνομαι πως διέπραξα τεράστιο σφάλμα. Θα έπρεπε να ξεκινήσω την παρουσίασή μου πρώτα απ' όλα με το θέμα της προστασίας IPR για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως αυτό να διατηρούσε το ενδιαφέρον των συναδέλφων δεδομένου και της προηγούμενης συζήτησης. Επίσης θα συμφωνήσω με τον κύριο Σούστα, τον συνάδελφο, για την ιδέα για καλύτερη για καλύτερους κανόνες και δεσμευτικούς κανόνες. Γιατί μπορούμε να το πράξουμε αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε τις συνθήκες δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Και επίσης, προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη-μέλη δεν δεν είναι η μία ίδια με την άλλη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μάλιστα πολύ διαφορετικέ από τη μια χώρα στην άλλη. Άλλο είναι μικρομεσαία στη Βουλγαρία ή την Ρουμανία ή την Πολωνία και άλλο είναι μικρομεσαία στην Γερμανία ή την Σουηδία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε πάντοτε υπόψη. Χρειάζεται πρόσβαση στις αγορές και για την εσωτερική αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των νέων κρατών μελών. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Συστήσαμε λοιπόν τις απόψεις 25-26 Απριλίου για ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή. Κύριο Σλίτερ, στα διάφορα πρόεδρε, αφού κλείσει αυτό έχω κάτι. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Μια και θα ψηφίσουμε τώρα στις 3. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών για, ανάθεση, για τροποποίηση της ε, αποφάσεως ποια είναι. Καλώ. θα ζητήσω από τον εισηγητή να μας κάνει μια πρόταση. διότι αν κάνω εγώ την τροπολογία μου στα Σουηδικά θα είναι έτοιμη στη μετάφραση μέχρι, τα τρι, μέχρι τις τρεις; Ναι, ναι, όχι, μπορείτε, μπορείτε. κάνετε ό,τι νομίζετε. Καλώς και ευχαριστούμε τους διερμηνείς που έμειναν μαζί μας. Κάτι παραπάνω. Thank you